Νομίζω ότι καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε. Λυπούμε που δεν είναι και άλλα μέρη εδώ, αλλά έχουμε τον κύριο Κάμπο, την κυρία Σμιτ, την κυρία Βανιού. Η Μπερναντέτ θα καθίσει εδώ.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 να ακούσουμε την παρουσίαση μιας μελέτης to a payment. μιας μελέτης για το το βασικό λογαριασμό πληρωμής, πληρωμών η κυρία Γκέπχαρτ θα μας παρουσιάσει ως εισηγήτρια για το ίδιο θέμα τη μελέτη αυτή και από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε και την ακρόαση για το ίδιο θέμα για την πρόσβαση σε ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό ε, στις 4 η ώρα. Αλλά αρχίζουμε πρώτα με την παρουσίαση που σας έλεγα. Um, sorry, I uh, So um, we're very pleased to have uh, Mr. Patrice. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι εδώ ο Πάτρις Μούλερ που είναι από το London Economics που έχει κάνει μια σχετική μελέτη στο παρελθόν είναι γνωστό στο Κοινοβούλιο του ανετέθη η δουλειά για το θέμα των βασικών τραπεζικών υπηρεσιών και φαντάζομαι ότι έχετε στο φάκελ λόσας και τη μελέτη και τις διαφάνειες που θα μας δείξει. Τώρα να ρωτήσω την κυρία Γκέπχαρτ, ως εισηγήτρια θέλετε να κάνετε μια εισαγωγή ίσως. Ναι. Ευχαριστώ πρόεδρε δεν θα μπω στην ουσία του θέματος. Μετά την παρουσίαση της μελέτης θα πω μερικά πράγματα. Απλά θα ήθελα να υπενθυμίσω πως το θέμα αυτό είναι γνωστό. Τα προβλήματα που συνδέονται με το θέμα αυτό είναι σημαντικά προβλήματα για τους πολίτες και είναι γεγονός ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Χαρήκαμε ιδιαίτερα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα εργασίας 2012 ανήγγειλε ότι θα αναλάβει νομοθετικό έργο για το θέμα αυτό και για προβλήματα δηλαδή που συνδέονται με την δυνατότητα πρόσβασης σε ένα βασικό λογαριασμό αλλά τελικά απογοητευθήκαμε όταν πήραμε μία ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα ασχοληθούμε νομοθετικά με το ζήτημα είναι, δεν είναι ικανοποιητικό αυτό διότι ξέρουμε ότι πάρα πολλοί πλήττονται, φύγονται από αυτή την υπόθεση γύρω στα 30 εκατομμύρια ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα διαφορών κατηγοριών από τους σπουδαστές Εράσμους που σπουδάζουν σε μια άλλη χώρα και ξαφνικά δεν μπορούν να υπογράψουν ενοικιαστήριο συμβόλο δίχως τραπεζικό λογαριασμό και τραπεζικό λογαριασμό δεν μπορούν να ανοίξουν αν δεν έχουν συγκεκριμένη διεύθυνση κατοικίας. Υπάρχει και η άλλη κατηγορία που, ε, των ανθρώπων που είναι υπερχρεωμένοι, έχουν οικονομικά προβλήματα, είναι αφαιρέγγοι αν θέλετε, αλλά σε προσωπικό επίπεδο χάσανε τα πάντα. Ξέρουμε βεβαίως ότι στον κόσμο μας συμβαίνουν και αυτά και ξέρουμε όλοι μας σε τελευταία ανάλυση ότι κανείς δεν μπορεί να ζήσει την καθημερινότητά του δίχως ο τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται ο μισθό του, οι αμοιβέ του, από τον οποίο πληρώνεται το νίκη του κτλ. Γι' αυτό αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα αναλάβουμε την πρωτοβουλία, θα κάνουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για να πιέσουμε και με αυτόν τον τρόπο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με το ζήτημα ε, Φόσον δεν το έκανε το 2011 ας το κάνει το 2012 και εντωμεταξύ είπαμε ότι αναθέσαμε και μια μελέτη για το ζήτημα για να μπορέσουν να μελετηθούν οι διάφορες πτυχές του θέματος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο εμπεριστατωμένα. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που ο κύριος Μίλλερ είναι εδώ για να μας παρουσιάσει τη μελέτη αυτή και αργότερα στην ακρόαση να δούμε και με τους τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να φροντίσουμε οι πολίτες της Ευρώπης να μπορέσουν να βιώσουν τελικά στην πραγματικότητα τα δικαιώματα τα οποία έχουν ούτως ή άλλως. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή αυτή που κάνατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τον Φίλιπ Έλε, ο οποίος ε, είναι, ε, εργάζεται για την Κομισιόν στη Γενική Διεύθυνση ΜΑΤ και είναι τιματάρχης για τα θέματα ακριβώ αυτά. Ε, όπως σας είπα την ε, παρουσίαση για τη μελέτη θα μας την κάνει ο κύριο ο Πάτρις Μίλλον ο οποίος εργάζεται στην Αγγλία και το γνωρίζω και από την ε, Αγγλία βέβαια, όπως έλεγε και η Εύλιν Γκέπχαρτ είναι ε, πολλά τα προβλήματα που δημιουργούνται από την μη πρόσβαση τραπεζικό λογαριασμό ενώ η πρόσβαση αυτή είναι βασικό καθήκον των Ευρωπαίων πολιτών δικαίωμα με συγχωρείτε των Ευρωπαίων πολιτών Αν δεν μπορείτε να δείτε τη διαφάνεια στο διαδίκτυο, ειδοποιώ τους ακροατές μας ότι θα τις ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα μας αργότερα. Ο κύριος Μιούλερ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και την εισαγωγή σας. Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες της μελέτης, γιατί είναι πάρα πολλές και θα χάσουμε χρόνο έτσι. Πάντως θα ήθελα να σας συστήσω, αν είναι δυνατόν, να διαβάσετε την έκθεση και να δείτε τα δεδομένα που περιλαμβάνονται εκεί. Είναι αρκετά ενδιαφέροντα και σημαντικά. Λοιπόν, στη σημερινή παρουσίαση θα ξεκινήσω αναφέροντας τους στόχους της μελέτης. Θα σας δώσω μερικά βασικά στοιχεία. Θα μιλήσω για τη σύσταση την ευρωπαϊκή για πρόσφαση στις βασικές, ε, στο βασικό λογαριασμό πληρωμών. Μετά θα, δω, θα συζητήσω λίγο το ποιες θα πρέπει να είναι αυτές οι βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και τα ε, ωφέλη αυτών και μετά θα καταλήξω σε κάποιες συστάσεις. Για τους στόχους. Όπως ξέρετε όλοι, η πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες ε, ε, την σήμερα ημέρα είναι απαραίτητη για την καθημερινότητα όλων. Για, για να έχει κανείς και τη δυνατότητα να αγοράσει το διαδίκτυο, να, να ζήσει καθημερινά. Χρειάζονται όλα αυτά κάποιο τραπεζικό λογαριασμό. Γιατί, διότι η κοινωνία γίνεται πάβει να είναι κοινωνία χαρτιού κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχουν πολλές επιταγές, check αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιούνται. Ή τα εμβάσματα γίνονται ηλεκτρονικά, είτε στην τράπεζα είτε με... Ε, λογαρια... από τον ίδιο τον δικαιούχο του λογαριασμού στο ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στα 30 εκατομμύρια ενήλικες άνω των 18 ετών δεν έχουν πρόσβαση όμως σε τραπεζικό λογαριασμό. Είναι πάρα πολύ ψηλό το νούμερο αυτό. Είναι κακό για και για την κατανάλωση αυτό αν θέλετε διότι οι πολίτες αυτοί δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ε, ε, ε, οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται στα διάφορα κράτη-μέλη για την πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό πληρωσμό, πληρωμών. Θα σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή και θα σας δώσω και μερικά στοιχεία για τα ωφέλη τα οποία θα μπορούσαν να προέλθουν αν οι άνθρωποι αυτοί είχαν πρόσβαση σε βασικό τροπεζικό λογαριασμό. Τρίτο θέμα που έλεγα να αναφέρω αλλά τελικά δεν θα αναφέρω ε, είναι αυτό των τελών που επιβάλλουν οι τράπεζες για τις διάφορες υπηρεσίες τους. Δηλαδή τι κοστίζει να έχει κανείς πρόσβαση ε, σε λογαριασμό ή να έχει ένα τραπεζικό λογαριασμό. Υπάρχουν πάντως τα στοιχεία, θα τα, δεν θα αναφερθώ στο θέμα αυτό τώρα, αλλά θα δείτε ότι τα πράγματα, θα το δείτε τα στοιχεία στο παράτημα και θα δείτε ότι διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα και από χώρα σε χώρα. Αυτή τη στιγμή τώρα για την πρόσβαση ε, στις τραπεζικές υπηρεσίες. Ποια είναι η κατάσταση στις διάφορες χώρες. Σε 12 κράτη-μέλη υπάρχουν κάποια προαπαιτούμεν, υπάρχει δυνατότητα, προβλέπεται, να δίνεται κάποια μορφή λογαριασμού. Σε 15 όμως κράτη-μέλη δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις, ούτε νομικές ούτε άλλου είδους διατάξεις. Δεν υποχρεωμένες τράπεζες να παράσχουν ένα είδος λογαριασμού. Άρα στη μειοψηφία, στα λιγότερα κράτη-μέλη, λιγότερα από τα μισά κράτη-μέλη δίνουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε κάποιες χώρες ορίζεται νομοθετικά ή κανονιστικά η υποχρέωση αυτή να υπάρχει ένας βασικός λογαριασμός. Σε άλλες χώρες είναι εθελοντικοί οι κώδικες, δεν είναι νομοθετημένοι. Αλλά βεβαίως η πρόσβαση στο λογαριασμό και οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι διαφορετικές. Στη Γαλλία, Βέλγιο, Φινλανδία και Δανία έχει κανείς πρόσβαση σε ε, τραπεζικές υπηρεσίες που ε, η πρόσβαση αυτή δίνει τη δυνατότητα να κάνει κανείς ό,τι χρειάζεται σε γενικές γραμμές. Στη Σουηδία μπορεί κανείς να έχει λογαριασμό καταθέσεων αλλά δεν μπορεί κανείς να κάνει ηλεκτρονικές πληρωμές. Δηλαδή, αν θέλετε να αγοράσετε στο διαδίκτυο μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό στη Σουηδία. Στην Ολλανδία ε, έγινε διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατικών αρχών και των τραπεζών για το δικαίωμα αυτό. Κατέληξε η διαπραγμάτευση σε μια συμφωνία ε, η οποία είναι υποχρεωτική, το αποτέλεσμα της οποίας είναι, είναι υποχρεωτικό, σε άλλες χώρες όμως είναι εθελοντική η δυνατότητα πρόσβαση, κανόνες. Είναι εκούσιοι αν θέλετε. Υπάρχουν κανόνες όπου γίνονται έλεγχοι για την ε, νομιμοποίηση παρανόμων προσόδων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο κώδικας λέει ότι υπάρχουν ειδικοί βασικοί λογαριασμοί πληρωμών, δεν είναι οι κανονικοί. Στην Ιταλία λέγεται... Ε, οι τράπεζες από μόνες τους έχουν πει ότι δίνουν τη δυνατότητα να ανοίξει κανείς ένα λογαριασμό. Τώρα, βέβαια υπάρχουν και αποχρώσεις στη Γαλλία. Έχει κανείς δικαίωμα να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό, αλλά μπορείτε να πάτε σε μια τράπεζα και η τράπεζα να πει εγώ δεν ανοίγω λογαριασμό και στέλνει τις πληροφορίες για στην κεντρική τράπεζα, η τράπεζα της Γαλλίας και η κεντρική τράπεζα μετά σας βρίσκει τράπεζα εμπορική η οποία θα σας ανοίξει το λογαριασμό. Άρα τα πράγματα δεν είναι απλά ακόμη και σε εκείνες τις χώρες που έχουν νομοθετήσει ε, σχετικά. Και είναι και αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι πολλές οι κατηγορίες πολιτών που πλήττονται λόγω της μη ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού, αυτοί που είναι ιδιαίτερα κινητικοί που φεύγουν από τη χώρα τους και πάνε κάπου αλλού, ε, και η διαδικασία ε, πολλές φορές είναι ταλαιπωρία. Ταλαιπωρείται ο πολίτης μέχρι να ανοίξει το λογαριασμό. Πιστεύουμε ότι κάποια δυνατότητα πρέπει να υπάρχει για ένα βασικό λογαριασμό ε, και από εκεί και πέρα βέβαια οι λεπτομέρειες συζητιούνται. Το Ευρωβαρόμετρο το 2010 έκανε μια δημοσκόπηση στην οποία οποία ζητούσε από τους ερωτώμενους να πούν κατά πόσον δυσκολεύτηκαν να έχουν πρόσβαση σε ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Η ερώτηση είναι κατά πόσον αντιμετώπισαν δυσκολίες. Όχι αν ήταν δυνατό ή όχι. Άλλο είναι αυτό το ερώτημα. Τέλος πάντων, ακόμη και για τις δυσκολίες βλέπουμε ότι ε, από τις απαντήσεις στο Ευρωβαρόμετρο ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές 39% στη Ρουμανία είπαν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες 5% ή λιγότερο από 5% στη Φινλανδία και στην Ολλανδία αντιμετώπισαν δυσκολίες άρα τίθεται το ερώτημα υπάρχουν προβλήματα υπάρχουν φραγμοί υπάρχουν ε, ε, πράγματα εμπόδια τα οποία για να περιπηδηθούν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε κι εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να μπορέσουν να αρθούν οι φραγμοί αυτοί μιλάμε υπάρχουν βέβαια δεν υπάρχουν χώρες που δεν προβλέπουν πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Αλλά εκεί προβλέπονται ιδιαίτερα πολλές δυσκολίες σε κάποιες χώρες. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε μια ε, σύσταση για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, αυτή ουσιαστικά η αποτυχία της αγοράς. Γιατί είναι αποτυχία της αγοράς ε, τελικά. Και ποια είναι η αρχή. Η αρχή είναι ότι όλοι οι καταναλωτές που είναι νόμιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν, πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν και να χρησιμοποιούν ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αν δεν έχουν ήδη λογαριασμό σε αυτό το κράτος μέλος. Αυτή, η αρχή αυτή είναι ιδιαίτερα ευρεία. Ποιοι είναι οι στόχοι της. Δύο. Αφενός δεν πρέπει να ε, υπάρχει αποκλεισμό κάποιων κοινωνικών κατηγοριών στα οικονομικά, από την οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωσης ε, αυτή ε, και αυτό συνδέεται με την ύπαρξη της ενιαίας εσωτερικής αγοράς αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος στόχος τον οποίο θα το δούμε αργότερα τώρα για την Λέει η σύσταση επίσης ότι θα πρέπει ο βασικός τραπεζικός λογαριασμός ο οποίος ανοίγει να είναι δωρεάν ή να ευλόγου κόστους. Τώρα τι θα πει ευλόγο κόστο, είναι δύσκολο να οριστεί. Αν πάση περιπτώσει όμως ε, και λέγεται ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια εκστρατεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, συνειδητοποιήσουν τα κράτη-μέλη την υποχρέωση που έχουν. Βεβαίω τώρα λέμε υποχρέωση αλλά δεν υπάρχουν κυρώσει εάν κανείς δεν ε, ε, κάνει ε, δεν, δεν αναλάβει τη, αν κάποιο κράτος δεν αναλάβει τη δέσμευση αυτή. Τι να πούμε, το ερώτημα που τίθεται βέβαια είναι αν δεν κάνουν τίποτα τα κράτη-μέλη και το δούμε σε μερικά χρόνια τι θα γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε. Τα κράτη-μέλη θα έτουν εμπόδια στην ε, ενιαία εσωτερική αγορά. Τόσο απλά περιγράφεται αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Λοιπόν, τώρα, τι θα Τι υπηρεσίες πρέπει να παρέχει αυτός ο βασικός τραπεζικός λογαριασμός για να δούμε τι υπηρεσίες πρέπει να παράγονται. Ε, μελετήσαμε τη βιβλιογραφία από διάφορους οργανισμούς, ενδιαφερόμενους φορείς κτλ. Και υπάρχει μια, ε, όχι ομοφωνία, αλλά μεγάλη συνένεση ότι ο βασικός λογαριασμός θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, θα πρέπει να μπορεί το άτομο να ανοίξει, να διαχειριστεί και να κλείσει το λογαριασμό. Θα πρέπει να μπορεί να καταθέτει και να κάνει αναλήψεις. Κατάθεση και ανάληψη. Και πρέπει να επιτρέπει και πληρωμές μέσω είτε μέσω εμβασμάτων είτε μέσω κάποιας κάρτας, τραπεζικής κάρτας. Εδώ αρχίζουν να υπάρχουν τα προβλήματα. Γιατί, διότι αν μπαίνουν τα χρήματα στο λογαριασμό σας, αλλά μετά δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, τότε μοιραία περιορίζεται η συμμετοχή σας στην οικονομία. Και δεν είναι δυνατόν να μην μπορείτε να κάνετε εμβάσματα από τη μια τράπεζα στην άλλη ηλεκτρονικά ή να μπορείτε να κάνετε πληρωμές κλπ είναι πολύ σημαντικό οι υπηρεσίες αυτές ε, που παρέχονται από τις τράπεζες να μην είναι συνδεδεμένες, δηλαδή συνδεδεμένες με κάποιο τραπεζικό προϊόν κτλ. Να είναι τελείως αυτόνομες και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά. Τώρα, τι γίνεται με αυτούς που έχουν οικονομικές δυσκολίες. Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να ε, έχουν προβλήματα στη χείριση του λογαριασμού της, ε, να έχουν προβλήματα ρευστότητας κλπ. Δεν λέγεται βεβαίως ότι δεν μπορεί κανείς να να κάνει υπεραναλήψεις. Βάσει του λογαριασμού αυτού εδώ υπάρχει συνένεση, αλλά και, αυτό, και η υπερανάληψη γιατί απαγορεύεται, γιατί ε, δεν θα πρέπει ε, να εφόσον λέμε ότι δεν θα πρέπει να κοστίζει για αυτόν που ανοίγει το λογαριασμό, δεν θα πρέπει να κοστίζει και υπερβολικά για την τράπεζα μετά ο λογαριασμός αυτός. Λοιπόν, η σύσταση της Ένωσης είναι περιγράφει ακριβώς όλα αυτά ε, περιγράφει τις υπηρεσίες λοιπόν άνοιγμα, κλείσιμο και διαχείριση του λογαριασμού κατάθεση ε, ανάληψη, ανάληψη μετρητών και ε, δυνατότητα εμβασμάτων. Τώρα, τι εμβάσματα ε, δεν θα πρέπει, θα πρέπει να είναι άμεση ε, θα πρέπει να μην υπερβαίνει το όριο του περιεχομένου του τραπεζικού λογαριασμού το ποσό το οποίο τρα... αναλαμβάνεται, δεν υπάρχει υπερανάληψη, δεν μπορούν να δοθούν πιστοτικές κάρτες παρά μόνο χρεωστικές κάρτες. Αυτά όλα ε, είναι ε, σύμμορφα σύμφωνα με αυτά που προτείνουν και οι εμπειρογνώμονες του κλάδου. Άρα καλή η σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ωφέλη υπάρχουν. Εδώ κάποιο κόστος θα υπάρχει. Τι ωφέλη υπάρχουν όμως. Υπάρχουν ωφέλη για αυτούς οι οποίοι έχουν οικονομικές δυσκολίες, για α, τα άτομα εκείνα τα οποία κινούνται από τη μια χώρα στην άλλη θα υπάρχουν ωφέλη υπέρ του διασυνοριακού εμπορίου και του ηλεκτρονικού εμπορίου και τελικά θα υπάρχουν ωφέλη για την, κοινο... για κοινωνία. Να τα περιγράψουμε αυτά τα ωφέλη ε, λιγάκι γιατί ορισμένα πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα αλλά δεν είναι υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι, οι ε, ε, ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες αν παραδείγματο όταν δεν έχουν λογαριασμό δεν μπορούν να πιάσουν μια δουλειά γιατί δεν μπορεί να μπει πουθενά ο μισθός τους δεν, ε, δεν μπορούν να νοικιάσουν κατοικία διότι το νίκη περνάει την σήμερα ημέρα από την τράπεζα δεν μπορούν να πάρουν κοινωνικά επιδόματα τα οποία τους οφείλονται διότι δεν υπάρχουν επιταγές πια δεν πληρώνονται με τσεκ τα επιδόματα αυτά πάνε κατευθείαν σε κάποιο λογαριασμό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν άλλους ε, ε, τρίτους μέσω των οποίων να στείλουν ε, χρήματα σε κάποιον που θέλουν να στείλουν πάνε ε, στα γραφεία, τα ανταλλακτήρια ε, περνάνε από κάποια ανταλλακτήρια τα οποία τους κοστίζουν περισσότερο ενώ αν, ναι, έχει κανείς ε, μια τράπεζα ε, ένα τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να δώσει μια μόνιμη εντολή η οποία είναι πολύ φτηνότερη άρα και εδώ φορολογούμε τη φτώχεια αν θέλετε δίχως τον τραπεζικό λογαριασμό επίσης ε, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ηλεκτρονικές πληρωμές την χάνουν εκπτώσεων ε, υπάρχει πρόβλημα Υπάρχει πρόβλημα με την διακίνηση μεγάλων ποσών, αν δεν υπάρχει λογαριασμός. Ε, υπάρχει, και υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο διαδίκτυο σημαίνει πρόσβαση και για κάποια προϊόντα τα οποία πουλούν, πουλούνται φθηνότερα στο διαδίκτυο από ότι στο κατάστημα ή αλλού. Άρα λοιπόν αν δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και εκεί φορολογούμε τη φτώχεια και τελικά ε, υπάρχουν και ψυχολογικοί παράγοντες που παίζουν στην όλη υπόθεση η ύπαρξη το να έχει κανείς έναν τραπεζικό λογαριασμό σου δίνει άλλη αίσθηση άμα δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό θεωρείς ότι είσαι αποκλεισμένος από την κοινωνία και από την οικονομία. Αν ε, εξετάσουμε τώρα τα ωφέλη από τους ε, ε σε ό,τι φορά τη γεννητικότητα των ατόμων, το θέμα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να ανοίξει κανείς τραπεζικό λογαριασμό όταν έχει μόλις μετακομίσει από ένα κράτο μέλο σε ένα άλλο. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό είναι ότι διαφορετικού τύπου προβλήματος. Ενώ το θέματα ε, της μη ε, δημιουργίας τραπεζικού λογαριασμού πρόκειται από τα χαρακτηριστικά τη ε, ζήτησης, της, της το θέμα της κινητικότητας ε, των ατόμων, το πρόβλημα προκύπτει από τον τομέα της προσφοράς. Δηλαδή, η πλευρά της ε, προσφοράς δημιουργεί προβλήματα στα άτομα. Δεν είναι τα άτομα που έχουν πρόβλημα, γιατί θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Ξέρουμε ότι σε σημερινά περιπτώσεων οι, κινητικοί ε, πολίτες έχουν συγκεκριμένα προβλήματα, δυσκολία στο να χορηγήσουν κάποιο πιστοποιητικό ε, ή αν θέλετε κάποιο τύπο ταυτότητας του ατόμου. Υπάρχουν χώρες όπου ο μετανάστης ο οποίος έχει μόλι δεν έχει καν ταυτότητα μαζί του. Έχει παρατηρηθεί σε σειρά περιπτώσεων ότι οι νομικές απαιτήσεις που συνδέονται με τα θέματα απάτης ε, και καταπολέμησης ξεπλήματος ρόμικου χρήματος, ορισμένες φορές ερμηνεύεται από κάποιες τράπεζες με πάρα πολύ περιορισμένο τρόπο που και τους δίνει δυνατότητα ορισμένε φορές να κλείσουν τους λογαριασμούς ατόμων που μετακινούνται από μία χώρα σε, μία άλλη του κράτους, σε ένα άλλο κράτος μέλος. Ιδιαίτερα όταν ο πελάτης δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικός εμπορικά. Υπό την έννοια δηλαδή ότι έχουν προσδοκίες. Αν είσαι φοιτητή, ο λογαριασμό θα είναι πάρα πολύ μικρό, θα έχει πάρα πολλέ πληρωμέ και διακινήσει μέσα έξω και επομένω όλη αυτή η ροή προμηθειών για την τράπεζα μην είναι πολύ υψηλή. Σε αυτή την περίπτωση όπου υπάρχουν απαιτήσει καθεαυτές από την τράπεζα που χρησιμοποιούνται ή ίσως χρησιμοποιούνται και καταχρηστικά για να εμποδίσουν την πρόσβαση στο άνοιγμα ενός προσωπικού λογαριασμού. Το 2011, η μελέτη Ευρωβαρόμη του 2011 που ε, έκανε μια δημοσκόπηση μεταξύ των πολιτών για να δουν ποια ε, εμπόδια θεωρούν στην ενιαία εσωτερική αγορά, το άνοιγμα ενός προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού εντοπίστηκε και χαρακτηρίστηκε σε ένα από τα μείζωνα ζητήματα. Το να απαλλαγούμε λοιπόν από αυτό το πρόβλημα έλλειψης πρόσβασης σε τραπεζικό λογαριασμό για τους κινητικούς ε, καταναλωτές θα ενισχύσει την ενιαία αγορά. Γιατί είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι δυσκολεύονται στην κινητικότητά τους λόγω αυτού του, λόγου συγκεκριμένου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το διασυνοριακό και ηλεκτρονικό εμπόριο. Η, πιο πρόσφατη μελέτη της Eurostat σε ό,τι αφορά τις καταναλωτικές συνήθειες απέδειξαν ότι 12% εκείνων που δεν χρησιμοποιούν το ίντερνετ για να παραγγείλουν online ε, υπηρεσίες ε, ή εμπορεύματα σε σχέση με την 12μηνη περίοδο που, ε, που προηγήθηκε μιας άλλης πρόσφατης μελέτης Eurostat εμφανίζουν ακριβώς την έλλειψη προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού ή σχετικής κάρτας για αυτό το λόγο. Ένα από τα προβλήματα δηλαδή και ένα από τους λόγους που κάνουν ηλεκτρονικό εμπόριο είναι αυτό. Στην, η διαθεσιμότητα ε, πιστοτικών καρτών και ηλεκτρονικού χρήματος, αν θέλετε, μέσω άλλων ε, διάβλων είναι βασικοί παράγοντες για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδιαίτερα καθώς προσφέρουν στον καταναλωτή προστασία και, ε, ε, και αξιοπιστία. Γιατί μιλάμε το ηλεκτρονικό εμπορίο, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα κυρίαρχο διάβλος μέσω του οποίου οι καταναλωτές μπορούν να έχουν ε, ε, εμπορεύματα σε χαμηλή τιμή, αλλά επίση γιατί μπορούν να κάνουν αγορές διασυνοριακές. Υπάρχουν πάρα πολλοί διασυνοριακοί ε, συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Αλλά αν είναι να βγει κανείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οποιοδήποτε λοιπόν φραγμός στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ε, τη ευρία έννοια, ε, αναχαιτίζει, μπλοκάρει τον δρόμο προς την ενιαία εσωτερική αγορά. Συνοπτικά λοιπόν αυτά είναι τα μεγάλα ωφέλη τα οποία προκύπτουν εάν οι άνθρωποι έχουν σωστά και επαρκώς προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό σε, χώρες, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι συστάσεις. Είδαμε ότι τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού, έτσι όπως μας δόθηκε, αν θέλετε, τα βασικά χαρακτηριστικά, ε, συνάδουν με αυτές τις συστάσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν εφαρμοζόταν σωστά οι οδηγίες στα όλα τα κράτη-μέλη, κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση, τότε θα υπήρχαν πάρα πολλά ωφέλη και για τα άτομα τα οποία δεν έχουν δεσμευθεί ή δεν έχουν συνδεθεί με μια συγκεκριμένη τράπεζα ε, για να είναι πολύ πιο κινητικά και να, έχουν και να, να μετέχουν και εμπόριο. Αυτό που φοβόμαστε ότι ενδεχομένω ε, η σύσταση αυτή να μην ακολουθηθεί από πραγματική πολιτική σε επίπεδο εθνικού κράτους μέλους, δεν υπάρχει συνεργατική υποχρέωση. Θα ήταν λοιπόν ε, πρόσφορο σε κανένα δύο χρόνια να ξαναγίνει πάλι μια απογραφή της κατάστασης και να δούμε τι έχει αλλάξει, κατά πόσον τα, ε, ε, τα επιθυμητά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί. Εάν δεν έχει υπάρξει σχετική πρόοδο ή είναι απειροελάχιστη, εάν ο αριθμό των ατόμων που δεν συνδεμένα με τράπεζα εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό, κατά την άποψή μα θα έπρεπε να σκεφτούμε κάποια οδηγία που θα διασφάλιζε την, το θα της νομοθεσίας. Επειδή όμως τα τραπεζικά συστήματα ποικίλουν κατά κόρον στην Ευρώπη, οι πρακτικές, οι οργανισμοί, η οργάνωση των τραπεζών, ίσως θα ήταν καλό να σκεφτούμε μια οδηγία με, κάποιες ελάχιστες, ε, με κάποια ελάχιστη εναρμόνιση του τρόπου λειτουργίας ε, των τραπεζών, δίνοντας όμως ανοιχτό το επίπεδο στο πώ θα παρέχονται υπηρεσίε. Τη διακριτική, δηλαδή, ε, αφήνοντα δηλαδή στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Αυτά σας δίνω σε γενική σύνοψη. Υπάρχουν και περισσότερες πληροφορίες με την έκθεση, αλλά κλείνω εδώ για να έχουμε και λίγο χρόνο για συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, πολύ ευρύ αυτή παρουσίαση και ήταν μια πάρα πολύ δυσδετική μελέτη όσον αφορά τα ωφέλη αν υπάρχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Και το επεκτείνεται κιόλας ε, αυτό εξετάζοντας και πέραν των, ε, και συμπεριλαμβάνοντας και αναφέροντας και τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Η Επιτροπή αυτή σίγουρα θα μελετήσει παιδεία που, που ε, σε ό,τι αφορά τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κινητικοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπατε ότι πολύ σωστά υπάρχει, υπάρχει ο φαύλος κύκλος εάν θέλετε η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα σε σχέση με κάποιον ο οποίος θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι έχοντας έχος ε, μετακινηθεί από άλλο κράτος μέλος και ταυτόχρονα και ως εχέγγυο να είναι η, το, η ύπαρξη προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κατάλογο των αγοριτών. Θα έχουμε την ευκαιρία για ε, μία σειρά ερωτήσεων. Κυρία Γκέπχαρτ, θέλετε να ξεκινήσετε. Και μετά ο κύριος Σμιτ κυρία Τούρναν, ο κύριος Δεκάμπος, ο κύριος Κοφεράτη. Κανείς άλλος? Ωραία, ξεκινάμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιούλερ. Πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μας δώσατε. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε έτσι παρουσιασμένα πολύ συνεκτικά τα πράγματα, ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι πιθανές λύσεις, τι ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αυτά που είπατε επιρρονίουν την άποψή μου ότι η πρόσβαση σε ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό είναι ουσιαστικά καθολική υπηρεσία. Καθολική υπηρεσία η οποία πρέπει να είναι στη διάθεση όλων των ανθρώπων. Ξέρω ο, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν τραπεζικό λογαριασμό. εντάξει, αυτούς δεν θέλω να τους πιέσω. Άμα θέλουν να έχουν κάτω από το πάπλωμα τα λεφτά τους οι άνθρωποι, ας το κάνουν. Αλλά να, τουλάχιστον αυτοί που θέλουν να έχουν... Ε, ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα λογαριασμό. Α, βεβαίως όλα ε, αυτά εξαρτώνται και από το από το πώς δρούν οι διάφορες κοινωνίες από την, το αν θέλουμε να προωθήσουμε ή όχι το ηλεκτρονικό εμπόριο το διασυνοριακό εμπόριο κτλ, κτλ. πράγματα που θέλουμε να κάνουμε η, ο, οι συνθήκες βέβαια στα κράτη-μέλη ε, είναι, ε, οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές και το γιατί 39-40% των ανθρώπων στη Ρουμανία δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό δεν ξέρω ε, ίσως ε, δεν υπάρχουν τραπεζικοί ε, οργανισμοί, πολλά τραπεζικά ιδρύματα, ε, οι μικροπολιτές, ε, ο Μανάβης, ο Μπακάλης δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. <laughs> το ή ο μισθό δίνεται σε χαρτοσακούλα. Τι να σας πω, αν υπάρχουν τέτοια πράγματα, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε βεβαίως, αλλά ε, μπορεί κανείς να πάει από το ένα κράτος στο μέλος στο άλλο και με αυτή την έννοια να πάει σε ένα κράτος που δεν δίνει το μισθό σε σακούλα και να έχει πρόσβαση σε ένα τραπεζικό λογαριασμό εκεί αυτό μπορούμε να το ρυθμίσουμε υπάρχουν ε, λοιπόν προβλήματα είδαμε επίσης στη, στις διάφορες χώρες και στην ε, πολύ προηγμένη Φινλανδία αλλά και στη Βουλή. Βουλγαρία και στην ε, Ρουμανία. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα ιδρύματα στις διάφορες χώρες. Θα ήθελα να, να σας ρωτήσω αν αυτό το μελετήσατε, γιατί αυτό ίσως είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συγκεντρώσουμε όλες τις ερωτήσεις και μετά θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή για να απαντήσει. Κύριε Σμιντ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση της έκθεσης αυτής. Ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με όλα όσα ελέγχθησαν. Έχω μια κόρη η οποία σπουδάζει στο Ενδιμβούργο της Σκοτίας, που είναι μάλλον μια πολιτισμένη χώρα. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει να ανοίξει προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό. Έπρεπε να την βοηθήσουμε, να, να της δώσουμε εμείς, να είμαστε εμείς τριτεγγυητές κλπ. Εν πάση πτώση, με τις συστάσεις που βλέπουμε εδώ, γιατί βάζατε στο τέλος το, την ρήτρα, αν θέλετε, που είναι η πλέον σημαντική. Θα πρέπει να σκεφτούμε το θέμα των νομοθεσία. Συμφωνώ δηλαδή με τον εισηγητή ότι σε αυτό το νέο περιβάλλον αυτό είναι ένα βασικό εργαλείο για κάθε πελάτη, για κάθε συγγνώμη πολίτη να έχει τραπεζικό λογαριασμό. Και γιατί να περιμένουμε και να μείνουμε μόνο σε συστάσεις το 2012. Θα αντέστρεφα το επιχείρημα και θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε άμεσα την κατάλληλη νομοθεσία. Δεν είμαι τόσο υπέρ της κοινοτική νομοθεσίας, η πάγια θέση μου είναι αυτή. Αλλά αν τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να χειριστούν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό, πρέπει να το κάνουμε εμεί. Και αναφερόμένο. και σε αυτά που είπε ο Πιαμόντε, αυτό ακριβώ ήταν να πω. Ευχαριστούμε κύριε Τέντρο. Ευχαριστώ για την παρουσίαση ήταν ενδιαφέρουσα και υποστήριξε αυτά τα οποία έχει υπόψη της η Επιτροπή αυτή. Συμφωνώ μου από τον προηγούμενο μιλητή ότι ίσως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο τολμήροι στα βήματά μας. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο 15% του ευρωπαϊκού πληθυσμού που ένα 15% του ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει δυσκολία να ανοίξει προσωπικό λογαριασμό. Παρά υψηλό το ποσοστό, θεωρώ του 2012. Γι' αυτό ίσως αυτή η Επιτροπή θα μπορούσε να κινήσει τα πράγματα, να κινηθούν λίγο πιο γρήγορα. Το ερώτημά μου είναι πώς το ζωστό σχέδιο θα μπορούσε να λειτουργήσει στην πράξη. Γιατί είπατε στη Γαλλία, αν πας σε μια τράπεζα, ενδεχομένω σε απορρίψει και πρέπει να πας στην κεντρική τράπεζα και να ζητήσεις πληροφορίες, ε, συμβουλές, βοηθή, οτιδήποτε. Αυτό είναι θέμα και πολλοί θα εγκατέλειπαν την προσπάθεια αν μετά από δύο-τρεις απορρίψεις από δύο-τρεις διαφορετικές τράπεζες. Είναι λοιπόν δυνατόν να έχουμε νομοθεσία που θα καθιστούν αδύνατη την απόρριψη κάποιου πολίτη από κάποια τράπεζα. Είναι κομμάτι του μοντέλου σε κάποια χώρα σήμερα. Θα ήταν νομικά αδύνατον. Δεν μιλάω για να χορηγούνται δάνεια στα άτομα ή να έχουν όριο υπερανάληψης, αλλά να υπάρχει ένας βασικός ε, προσωπικός, ε, προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός, νομίζω είναι απόλυτα σωστό και δίκαιο. Κύριε Κάμπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την παρουσίαση αυτή. αλλά μου γέννησε και πάρα πολλές αμφιβολίες για να είμαι ειλικρινής. Κάθε μέτρο έχει και την αντίστροφη πλευρά. Ας δούμε το θέμα με τους σπουδαστέ. Αν περιορίσουμε τον τραπεζικό λογαριασμό των φοιτητών απλώς και μόνο σε αυτό που δεν του επιτρέπεται να έχουν μια πίστη, να τους χορηγείται κάποια πιστοτική γραμμή, τότε είναι, για, είναι δωρονάδρον, γιατί σε αρκετές στιγμές της ζωής θα χρειάζονται και κάποια σχετική, κάποιο σχετικό μικρό δάνειο ή κάποιο όριο, κάποια υπερανάληψη. Καταλαβαίνω βέβαια ότι πρέπει να το περιορίσουμε αυτό, αλλά κάθε μέτρο έχει και το αντίστροφό του. Ένα πεδίο όπου νομίζω ότι η εναρμόνιση θα έπρεπε να ακολουθήσει δύο πεδία. Το ένα είναι ε, ε, εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών από το σπίτι, που είναι πολλών παραλλαγών. Σήμερα, για παράδειγμα, σε αυτή τη χώρα που ζούμε τώρα, οι τραπεζικές αλλαγές από το σπίτι προϋποθέτει ειδικό εξοπλισμό που νοικιάζεις ή αγοράζεις για να μπορείς να έχεις πρόσφατο τραπεζικό λογαριασμό. Για να κάνεις μια ε, τραμεταβίβαση χρημάτων από ένα οργανισμό σε άλλον, πληρώνει πάρα πολύ ακριβά, γιατί δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει από το σπίτι, πρέπει να πα στο κισέ και ούτω καθεξή. Κατανοώ επίση ότι η διάθεση πιστοτικών καρτών, αυτή η επανάσταση που όλοι ζήσαμε στην αρχή της δεκαετίας του ήταν και ένας εκπληκτικός λόγος για την ε, αύξηση, κατακόρυφη και αύξηση των δανείων και που μας βήθησε στην τρέχουσα κρίση. Επομένως πρέπει να μελετήσουμε κάθε προτινόμενη σύσταση, κάθε μέτρο έχει και την αντίστροφη πλευρά του. Δεν θέλω να εμποδίσω με αυτά που λέω όσα προτάθηκαν, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη πάρα πολλά στοιχεία. Από αυτές τις στάσεις λέει και τα προτινόμενα κάποια μπορούν να είναι χρήσιμα και κάποια μπορούν να είναι παρακινδευμένα. Ευχαριστώ. Έχουμε δύο ακόμα ομιλητές. Πρωτού ζητήσω από τον κύριο Μίλερ να δευτερολογήσει. Ο κύριος Κοφεράτη καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ ότι εξεπλάγει όχι τόσο από την παρουσίαση, αλλά περισσότερο από τα διαγράμματα που καθιστούν ακόμα πιο εύγλωτα, εύγλωτη την ομιλία που παρακολούθησα εδώ πέρα από τον εισήγητη, από τον καθηγητή Μίλλερ. Αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι μια, ένα μεγάλο κομμάτι των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχουν αντικειμενικά, ε, δεν απολαμβάνουν αντικειμενικά ενός δικαιώματός τους. Είναι μια απουσία που απορρέει από πάρα πολλούς λόγους, ακόμα και παράγοντες ιστορικού χαρακτήρα, αλλά που θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη στην εποχή μας, στην αρχή της τρίτης χιλιετίας. Διότι το να μην έχουν πρόσβαση σε έναν ε, λογαριασμό, βασικό λογαριασμό όψεως, προκαλεί αναφυσβήτητα ένα πολύ μεγάλο περιορισμό στην, στην αγοραστική ικανότητα και επιλογής ε, των καταναλώσεων της οποιασδήποτε κατανάλωσης σε εκατομμύρια πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ' εμέ, είναι ένα δικαίωμα μη εγγυημένο ακόμα, με δεδομένο ότι για τόσους πολλούς εκατομμύρια ανθρώπους είναι εκτός. Πρέπει να βρούμε γρήγορη λοιπόν και αποτελεσματική λύση. Και σε μένα λοιπόν φαίνεται και θεωρώ ότι είναι σημαντικό υπό αυτές τις συνθήκες να σκεφτούμε με βάση κάποιο νόμο, όχι αφήνοντας στα μεμονωμένα κράτη-μέλη τη διακριτική ευχέρεια και το καθήκον αντιδράσεων. Γιατί η δράση των μεμονωμένων κρατών μας οδηγεί και πάλι στο πλαίσιο και στην κατάσταση που περιγράφεται ε, εδώ και που είσαι μέχρι σήμερα. Τα ιστογράμματα που βλέπουμε από την ε, εισήγηση του επιβεβαιώνουν. Είναι ένα είδος, αν θέλετε, προτεραιοτήτων που πρέπει να δούμε για να, γίν για εγγυηθούμε τα δικαιώματα όλων. Και το πιο αποτελεσματικό εργαλείο γι' αυτό είναι ακριβώς ένας ε, νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια μπορούν να προκύψουν στοιχεία προσαρμογής, απαραίτητης προσαρμογής στην εφαρμογή του νόμου αυτού και επί τη βάση των επιπτώσεων που παρέχει. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα το οποίο αφορά στη γνώση στη γνώση του υφιστάμενου πλαισίου και των υφιστάμενων μηχανισμών. Υπάρχει δηλαδή και μια διαδικασία εκπαιδευτική που θα πρέπει να υπάρξει για να παρουσιάσει τα διάφορα θέματα στον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Θέλω να κάνω μια ακόμα παρατήρηση στην ενισχυτική κατάσταση που περιγράφεται στην εισήγηση. Η σχεδόν υποχρεωτική χρήση των χρημάτων, του ρευστού δηλαδή, είναι μία από τις συνθήκες που πρημοδοτεί την διεύρυνση της ε, εγκληματικότητας, τα φαινόμενα εγκληματικότητας και διαφθοράς, ξεκινώντας από την ε, διαφθορά πολιτικών, βασίζεται ακριβώς διαθεσιμότητα των, του ρευστού χρήματος. Υπάρχουν λοιπόν αντικειμενικές ε, περιπτώσεις και επομένως διακινδυνεύεται ε, ασυνείδητα να η ευνόηση και η πρόθεση της εγκληματικότητας. Επομένως, η το δικαίωμα των ατόμων να έχουν στο τραπεζικό λογαριασμό, αλλά και να είναι απρόσκοπτη καθημερινή του ζωή. Κυρία Πέντεκοστ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ομιλητή για την εξαιρετική παρουσίαση. Ένα σύντομο ερώτημα έχω να υποβάλω. Θα ήθελα να το ρωτήσω αν υπήρξε προηγούμενη δουλειά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω στα εθελοντικά μέτρα και ποιο ήταν το αποτέλεσμα σε επίπεδο κρατών μελών. Και στην περίπτωση της αποτυχίας αγοράς η νομοθεσία είναι σωστός τρόπος να κινηθούμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική πρωτοβουλία και οφείλουμε πάρα πολλά σε εκατομμύρια άτομα. 30 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό είναι τεράστιο μειονέκτημα. Αν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στο ερώτημα αυτό, θα χαιρόμουν ιδιαίτερα. Και ευχαριστώ. Well, the... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ βρήκα πάρα πολύ ε, ευχάριστη την, ε, και επικοδομητική την παρουσίαση. Και για έναν άλλο λόγο, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλος συσχετισμός του ποσοστού ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση και κάποιων ε, θεσμικών συμφωνιών. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι ο κύριος Φόρμαν και ο κύριος Κλούτς, ο οποίος είναι ε, ο εισηγητής της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του θέματος, θα συμφωνήσει ίσως να περιλαμβάνεται στις λεπτομέρειες της έκθεσης. Αλλά το πιο ενδιαφέρον, αν έχω ε, ε, ε, σωστά αποκωδικοποιώ τα θέματα, είναι ότι η Εστονία που δεν έχει ούτε οικειοθελείς, ούτε θεσμικές αναγκαστικές συμφωνίες είναι μία από τις τρεις ε, κορυφαίες χώρες στην χρήση των διατραπεζικών συναλλαγών μέσα από το σπίτι. Βέβαια είναι και η χώρα που έχει το υψηλότερο ποσοστό ψηφιακά εγγράμματων. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ότι τα στοιχεία αυτά κατά πόσον με πείθουν ότι ένα επίσημο κοινοτικό νομοθετικό κείμενο θα μπορούσε να είναι η απάντηση. Ιδιαίτερα παρατηρώντας ότι στις κάτω χώρες όπου το δικαίωμα τραπεζικού ε, λογαριασμού προκύπτει από μια συμφωνία μεταξύ των αρχών και των ε, τραπεζών, επομένως είναι κάτι το επίσημο, ε, έχει επηρεάσει το υψηλό ποσοστό, στον πολύ υψηλό αριθμό ατόμων που έχουν πρόσβαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση του εισηγητή ως προς τις διαφορετικές τραπεζικές δομές και την περιπλοκότητα όλου αυτού του θύματος. Δεν μελετήσαμε πώς συνδέεται αυτό με τη δομή του τραπεζικού συστήματος γιατί δεν είχαμε αρκετό χρόνο. Έπρεπε να ολοκληρώσουμε τη μελέτη μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική προθεσμία. Ωστόσο, θα ήθελα να πω το εξής. Σε ορισμένες χώρες, και είναι κάτι που έχω δει εγώ ο ίδιος προσωπικά, δεν υπάρχει τραπεζική υποδομή στα χωριά. Και έτσι οι τράπεζες στέλνουν άτομα τα οποία ε, κάνουν το γύρο μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα και προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ινδία αυτή τη στιγμή, όπου μόνο στα χωριά ε, ο κόσμος μπορεί να έχει πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πιο καινοτόμες λύσεις. Δεν είναι όμως δυνατό να προσφέρουμε τραπεζικές υπηρεσίες σε κάποιους που ζουν σε περιοχές που δεν έχουν τέτοιου είδους υποδομές. Να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας, να βγούμε από την πεπατημένη, αυτό που ονομάζουμε να σκεφτούμε έξω από το συγκεκριμένο πλαίσιο για να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτό κατά πρώτο λόγο. Κατά δεύτερο λόγο, γιατί υλοποιήσαμε μία σύσταση, την εφαρμόσαμε, η οποία τελικά αποδείχθηκε αδύναμη. Ίσως εν γέννη είμαι αισιόδοξη προσωπικότητα, πάντοτε όμως ήθελα και θέλαμε να δούμε πώς θα την αξιοποιήσουν τη σύσταση αυτή τα κράτη-μέλη, προτού αποφασίζουμε ότι όντως χρειάζεται κανονισμός, ο οποίος φυσικά έχει υποχρεωτική ισχύ. Εσείς θα αποφασίσετε τι ακριβώς πρέπει να επιλέξετε. Αξίζει όμως τον κόπο να σκεφτεί κανείς ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει διάφορες προσεγγίσεις με περισσότερη ή λιγότερη επιτυχία. Αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος είναι πολύ σημαντικό. Στη Γαλλία νομοθετείται αυτό το θέμα, αλλά είναι περίπλοκη η άγουσα. Στην Ολλανδία και στην Αγγλία είναι πιο εύκολα τα πράγματα που δεν νομοθετείται δεν είναι σαφές ότι ένας κανονισμός θα λύσει όλα τα προβλήματα. Βεβαίως όμως και όντως υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να λυθούν. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Τίθεται και το ερώτημα των αντισταθμιστικών μέτρων. Μήπως είναι πολύ περιοριστικό το πεδίο των υπηρεσιών που, προσφέρ, που προτείνουμε. Ε, λέγεται ότι θα πρέπει να δίδεται και πίστοση σε συγκεκριμένους, δυνατότητα επίσταση σε συγκεκριμένους λογαριασμούς, να μιλούμε για ηλεκτρονική τραπεζική και το καθεξής. Νομίζω ότι ξεπερνάνε όλα αυτά ε, το πεδίο εφαρμογής. Εδώ μας ενδιαφέρουν τα άτομα που έχουν ένα βασικό ε, τραπεζικό πρόβλημα. Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά και μπορείτε να τα προχωρήσετε ακόμα παραπέρα. Σε άλλο επίπεδο όμως. Από εκεί και πέρα έχουμε τις στατιστικές, τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου. Είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα. Ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες κατά πόσο δυσκολεύθηκαν να αποκτήσουν πρόσβαση, όχι κατά πόσο το θεώρησαν ανέφικτο το να αποκτήσουν πρόσβαση. Επομένως, κάποιοι από αυτούς που δυσκολεύτηκαν κατά πάσα πιθανότητα θα είχαν δει ότι ήταν αδύνατο να τελικά να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό. Το να έχεις δύσκολη πρόσβαση όμως δεν ισούται αυτομάτως με το να μην έχεις καθόλου πρόσβαση, να αποκλείεσαι από αυτή. Να μην εξάγουμε βιαστικά συμπεράσματα και να νομίζουμε ότι τελικά δεν απέκτησαν τραπεζικό λογαριασμό. Δεν συνεπάγεται αυτομάτως το ένα ε, το άλλο. Πέρα από αυτά, ε, τέθηκαν πολλές ερωτήσεις για το ποιος θα ήταν ο καλύτερος δρόμος να ακολουθήσουμε, μία οδηγία ή έναν κανονισμό. Απαντώ και πάλι λέγοντας ότι πρέπει πρώτα να δούμε αν σημειώνουν πρόοδο τελικά τα κράτη-μέλη και στη συνέχεια να δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες ποια θα είναι τα ωφέλη αλλά και τα μειονεκτήματα της κάθε μία προσέγγισης που υιοθετέ, υιοθέτησε η κάθε μία από τις χώρες. Και να διορθώσω κάτι αναφορικά με τη Γαλλία. Πριν από λίγα χρόνια πήγαινε σε μια τράπεζα και αν σου αρνεί η τράπεζα να σου ανοίξει λογαριασμό, μπορούσες να πας στην κεντρική τράπεζα της Γαλλίας αυτομάτως. Και τελικά ε, αυτό φάνηκε ότι δεν ήταν καθόλου λειτουργικό. Σήμερα έχει αλλάξει η νομοθεσία και οι διατάξεις προβλέπουν ότι η τράπεζα που αρνείται να ανοίξει λογαριασμό, οφείλει να διαβιβάσει τις πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα και η Κεντρική Τράπεζα θα στείλει την πληροφόρηση ε, στην άλλη τράπεζα η οποία έχει εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί ως τράπεζα που δίνεται να ανοίξει λογαριασμό στο άτομο. Δηλαδή εσείς ως άτομο δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα μπορεί κανείς να νιώσει κάποιο άγχος σκεπτόμενος ότι τα χαρτιά που με αφορούν τελικά θα καταλήξουν στην Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας, όμως τα πράγματα είναι καλύτερα σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι κατάφερα να απαντήσω ε, σε όλες τις ερωτήσεις και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα παραμένω στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε κύριε Μιούλερ, σας παρακαλώ να μείνετε μαζί μας για να συμβάλλετε περαιτέρω στη συζήτηση. Θα προχωρήσουμε ε, θα αφήσουμε τη δική σας παρουσίαση και θα περάσουμε στην ακρόαση. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους προσκεκλημένους και να πω ότι η Επιτροπή ανέθεσε στην London Economics να εκπονήσει μία μελέτη για τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Ε, αυτή η μελέτη περιλαμβάνει πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα στοιχεία για την τις τραπεζικές υπηρεσίες και την απουσία αυτών και πόσο αντίκτυπο έχει στη ζωή των συμπολιτών μας. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτή τη μελέτη από, την, από το διαδίκτυο και βεβαίως θα τη μοιράσουμε εδώ στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Τούτων λεχθέντων, θα ήθελα λοιπόν να κηρύξω επισήμως την έναρξη της δημόσιας ακρόασης να καλωσορίσω για άλλη μια φορά τους δύο εισηγητές, την κυρία Εύελιν Γκέμπχαρντ από την Επιτροπή της Ενίας Αγοράς και τον Γιούγκεν Κλούτερ από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Χαίρομαι ιδιαίτερος διότι έχουμε τον Τζόναθαν Φόλ εδώ μαζί μας, ε, Γενικό Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση για την ενίαγορα. Αγορά. Θα ήθελα να κάνω κάποιες αναρκτήριες παρατηρήσεις και στη συνέχεια ε, θα έχουμε δύο εμπειρογνώμονες που θα πάρουν το λόγο. Βασική τραπεζική ως δικαίωμα του καταναλωτή και καθελική υπηρεσία και πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών και ωφέλη για την ενιαία αγορά. Γι' αυτά θα μας μιλήσουν οι δύο εμπειρογνώμονες έχοντας ακούσει και τους εισηγητές πρώτα. Έχετε τα βιογραφικά στοιχεία των ομιλητών στο φυλάδιο που είναι διαθέσιμο στην αίθουσα. Δεν θα επεκταθώ να δώσω καταρχάς το λόγο στην Εύελιν και για να μας κάνει κάποιες εισαγωγικέ παρατηρήσεις. Μετά ο Γιούγκεν και μετά ο Τζόναθαν. Εύελιν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που οργανώθηκε η ακρόαση αυτή ακριβώς για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς πολίτες. 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση σε ε, βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Μιλάμε για άτομα άνω των 18 ετών και είναι πραγματικά διανόητο αυτό. Εγώ όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το θέμα δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός αυτών που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Λοιπόν, ε, άρχισα δεν άρχισα πέρσι να ασχολούμαι με το θέμα πέρσι. Εδώ και δέκα χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, έχει αρχίσει, άρχισε να συνειδητοποιεί ότι υπάρχει πρόβλημα και το 2008 ε, ξέδωσε μια σύσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύριος Μόντι όταν ήταν επίτροπος είπε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιηθεί στο θέμα αυτό. Είπε ο κύριος ε, έλεγε ο κύριος Μόντι ότι η Κομισιόν θα πρέπει να προτείνει ένα σχέδιο κανονισμού ε, το οποίο να προβλέπει για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ε, το δικαίωμα να έχουν να χρησιμοποιούν ε, κάποιες βασικές τραπεζικές υπηρεσίες για να μπορέσει να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολύ, εδώ και πολύ καιρό ε, τέθη το θέμα και το, ο Λούι Γκρέσ ασχολήθηκε εδώ στο Κοινοβούλιο τότε με το θέμα αυτό. Και ε, στο τέλος μας είπε η Κομισιόν ότι ναι, ε, θα προτείνει ένα σχέδιο οδηγίας. Όμως απογοητεύτηκα ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν έκανε τίποτα. Υπάρχει μια σύσταση της Κομισιόν όπως ε, ε, σας είπα, αλλά η σύσταση τι σημαίνει, ότι αν κάποιο κράτος μέλος δεν θέλει να κάνει κάτι τι, δεν είναι υποχρεωμένο να το κάνει. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια για να γίνει κάτι τι, όχι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό για τα 30 εκατομμύρια κόσμος, κόσμο που ζουν στην Ευρώπη και που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Αν κάποιοι βέβαια από αυτούς θέλουν να έχουν κάτω από το μαξιλάρι τους στο παπλωμά τους τα χρήματά τους, είναι δικαιωμά τους, μπορούν να το κάνουν. Απ' την άλλη μεριά όμως ε, αν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν ένα τραπεζικό λογαριασμό και δεν μπορούν να τον ανοίξουν, δεν έχουν πρόσβαση σε ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό, αυτό είναι αδιανόητο. Νομίζω ότι είναι δικαίωμα το. Πρέπει να πρόκειται για δικαίωμα των πολιτών να έχουν ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Την σήμερα ημέρα που ζούμε σε ένα ψηφιακό κόσμο πώς θα, πού θα μπει ο μισθός των ανθρώπων αυτών, πού η αμοιβή του, που θα, ε, πώς θα πληρώσει το νίκη του πώς θα αγοράσει κάτι στο ίντερνετ πώς θα λειτουργήσει τελικά η εσωτερική αγορά αν 30 εκατομμύρια πολίτες δεν έχουν λογαριασμό ε, εγώ ε, όταν πρώτο σκέφτηκα ότι θα κάνουμε μία ιδέα νομοθετική πρωτοβουλία έκθεση, ότι θα έπρεπε να το κάνουμε, όπω σα είπα δεν το περίμενα ότι είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι χωρίς λογαριασμό τραπεζικό και ότι τα συστήματα είναι ε, τόσο διαφορετικά στα κράτη-μέλη που δεν είναι λόγο θέλουμε εμείς να επιβάλλουμε κανόνες στις τράπεζες ή να νομοθετήσουμε ε, για να να υποχρεωθούν να κάνουν ορισμένα ε, πράγματα οι τράπεζες. Όχι, εμείς σαν Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες, οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες μπορούν να κινηθούν ελεύθερα και να απολαύσουν αν θέλετε την εσωτερική αγορά και με αυτή την έννοια να τονώσουν ή συμμετάσχουν στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένω λοιπόν ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μια γνωμοδότηση την οποία να πούμε και θα πω κάτι τώρα που είναι βαθιά πεποίθησή μου να πούμε ότι ε, χρειαζόμαστε νομική λύση η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί στα διάφορα κράτη-μέλη και να υποχρεώνει ουσιαστικά τα κράτη-μέλη να απαράσχουν ως δικαίωμα των πολιτών στους πολίτες την πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό. Έτσι ξεκίνησα τη δουλειά μου και χαίρομαι ιδιαίτερα που κάνουμε την ακρόαση αυτή σήμερα. Ε, έχουμε, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε και έναν συνάδελφο εδώ από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων είναι πολύ καλό αυτό και άσχετα βέβαια το ποια επιτροπή τελικά θα θεωρηθεί καθήλυνα αρμόδια ή όχι δεν με ενδιαφέρει νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτε μας να ζήσουν σωστά την καθημερινότητά τους στην κοινωνία της τρίτης χιλιετίας Ευχαριστώ ο, ο κύριος Κλούτ έχει το λόγο Ευχαριστώ πολύ Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω που με καλέσατε σήμερα εδώ Είμαι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων όπου πέρσι το Μάρτι κάναμε μια μόνη βέβαια μια ακρόαση για συναφή θέματα χαίρομαι λοιπόν που σήμερα μπορούμε και συναντιόμαστε εδώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτά που είπε η κυρία Γκέιπχαρτ ε, τώρα. Τι να... Πρόκειται για σοβαρότατο πρόβλημα. Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ε, βεβαίως υποστηρίζει και την επιβολή κανόνων στις τράπεζες ε, για άλλα θέματα αλλά σίγουρα για την πρόσβαση και το δικαίωμα των πολιτών να έχουν ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό δεν έχω τίποτα παραπάνω να πω εδώ ε, εκτός αυτή τη στιγμή ζούμε μια σοβαρή οικονομική κρίση και οι πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκαναν οι ίδιοι θυσίες έδωσαν και αρκετά λεφτά τελικά μέσω των κρατικών αρχών για να υποστηρίξουν τις τράπεζες. Ε, κάτι θα πρέπει, κάπως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και αυτοί τις τράπεζες. Κάτι θα πρέπει να κερδίσουν από τις τράπεζες ακούγεται και αυτό με αυτή την έννοια είναι και από πολιτικής απόψεως πολύ σημαντικό να ε, μάθει ο πολίτης τι προσπαθούμε να κάνουμε και από πολιτικής απόψεως να λύσουμε τα προβλήματα αυτών των 30 εκατομμυρίων πολιτών. Η και Κέιπχαρτ αναφέρθηκε σε παρα... στα προβλήματα, στους λόγους για τους οποίους δικαιολογείται η ανάληψη πρωτοβουλίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καθόλου καμία αντίρρηση από πλευράς δικής μας Επιτροπής ότι πρέπει να πρόκειται για νομοθετική πρωτοβουλία. τι να σας πω, να σας πω τι είπαμε στη συζήτηση που κάναμε στην Επιτροπή μας. Ίσως μία, ένα θέμα που είπαμε είναι ότι είναι γεγονός και διαπιστώνεται από όλου ότι οι συναλλαγές πολλές σε μετρητά δεν γίνονται πια οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται ε, ηλεκτρονικά και γι' αυτό θα πρέπει εφόσον θέλουμε να υποκαταστήσουμε αν θέλετε την, α, τις συναλλαγές με μετρητά με άλλου είδους συναλλαγές θα πρέπει κατά τη να είναι δωρεάν οι συναλλαγές αυτές βεβαίως η ηλεκτρονική συναλλαγή δεν μπορεί να μην έχει κανένα κόστος Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν συμπολίτε μας που δεν θέλουν να καταβάλουν το κόστος αυτό. Γι' αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να πούμε και να, δηλώ, και να καταστήσουμε σαφές ότι αν θέλουμε να ε, αντικαταστήσουμε την συναλλαγή με μετρητά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με συναλλαγές ηλεκτρονικές ή με κάρτες και τα λοιπά θα πρέπει να δώσουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα στους πολίτες όχι να είναι απολύτως δωρεάν αυτές οι συναλλαγές αν και ίσως θα έπρεπε να είναι δωρεάν ε, κατά τη δική μου άποψη αλλά τέλος πάντων ε, ας μην είναι δωρεάν αλλά τουλάχιστον να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις συναλλαγές οι πολίτες όλοι Άλλο θέμα. Ο βασικός λογαριασμός θα έπρεπε κατά την άποψή μας να προσφέρεται να προσφέρεται σε όλους ακόμα και αν δεν προσφέρει όλες βεβαίως τις ε, ε, ε, τραπεζικές υπηρεσίες. Δηλαδή, ακόμη και αν πρόκειται για έναν λογαριασμό ο οποίος ε, ουσιαστικά βασίζει, είναι λογαριασμός προνομών σε μετρητά που δεν επιτρέπει περαναλήψεις και τα λοιπά, θα πρέπει να προσφέρεται. Όμως, στην ακρόαση που κάναμε ε, πάρα πολλοί είπαν ότι τελικά η ύπαρξη ενός τραπεζικού λογαριασμού και η δυνατότητα υπερανάληψης ή δανεισμού κτλ. μέσω του λογαριασμού ε, είναι και ένα καλό εργαλείο για να μορφωθούν αν θέλετε για να εκπαιδευθούν συγγνώμη, οι νέοι ε, άνθρωποι, οι πολίτες της Ευρώπης σε θέματα διαχείρισης χρημάτων για να αποφευχθεί αύριο η υπερχρέωση παραδείγματος χάρη για να μπορούν να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα χρήματά τους επίσης για λόγους ανταγωνισμού ε, θα πρέπει να α, προσφέρουν τους λογαριασμούς αυτούς όλες οι τράπεζες. Φαντάζομαι ότι καμία τράπεζα δεν θέλει να μην προσφέρει κάτι που προσφέρουν όλες οι άλλες. Τώρα υπάρχει credit union και κάτι τέτοιου είδους ιδρύματα αν θέλετε ή ε, χρηματοπιστωτικά τα οποία μπορεί να είναι έξω από το τραπεζικό τομέα αλλά ε, στην Γερμανία να πω ότι παλιά δεν κάναμε τίποτα. Δεν γινόταν τίποτε στη Γερμανία. Ε, υπήρχε μια κάποια σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έκανε τίποτα η Γερμανία. Τώρα, μετά από μια εκστρατεία και μια, αν θέλετε, κινητοποίηση που έλεγε α, λογαριασμός για όλους, ε, για, λογαριασμός για τον καθένα, μετά από αυτή την κίνηση φαίνεται ότι οι τράπεζες ε, ε, άλλαξαν άποψη. Βεβαίως είπα, επιμένουν να έχουν... Ε, ε, επαφές με τον ε, υποψήφιο πελάτη και προσπαθούν ε, να μην δώσουν παράσχουν όλες τις υπηρεσίες και τα λοιπά όλα αυτά βέβαια το ότι υπάρχουν κενά με κάνουν να πιστεύω ακόμη περισσότερο ότι θέλει νομοθετική ρύθμιση το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ναι ναι τελειώνω στις 12 Μαρτίου θα συζητηθεί το πρώτο σχέδιο ο, της, μιας, της έκθεσης που θα φτιάξουμε μέχρι τις 25 περίπου 7 Απριλίου θα πρέπει μπορούν να κατατεθούν τροπολογίες και τα και το Μάη θέλουμε να κλείσει αυτή η υπόθεση να μπορέσουμε να ψηφίσουμε γιατί μέχρι την ε, ημερομηνία που μας έθεσε η Κομισιόν θα πρέπει να έχουμε κάτι έτοιμο να, ε, να δώσουμε. Αλλιώς δεν έχει νόημα το να κάνουμε χιλιάδες αναλύσεις και μελέτες και να μην μπορούμε τελικά να αντιμετωπίσουμε την Κομισιόν με, το, με κάτι απτό ε, για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια πολύ πιο ικανοποιητική ε, κοινή έκθεση. Τζόναθον Φόλ, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Να σου δώσω και σένα το λόγο για να μας πεις ε, ποια είναι η άποψη της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Μάλκομ. Αξιότιμα μέλη, κυρίε και κύριοι. Καλησπέρα σα. Να σα ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να παραστώ στην ακρόασή σας. Να σα ευχαριστήσω θερμά γιατί προτείνετε τη σύνταξη έκθεσης για το θέμα αυτό και εμείς περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να την διαβάσουμε την έκθεση αυτή. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι διακυβεύεται εδώ. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές όλο και περισσότερο αντικαθεστούν τις πληρωμές σε ρευστό για λόγους κόστους και ασφάλειας. Αλλά βεβαίως και για να διευκολύνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο όχι μόνο όχι μόνο διευκολύνουν, αλλά είναι και αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρχει ηλεκτρονικό εμπόριο. Εν πάση περιπτώσει, η πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία σήμερα, χωρίς να έχει κανείς τραπεζικό λογαριασμό, δεν είναι δυνατή. Καθημερινά πάμε όλο και προς μια κοινωνία η οποία θα κινείται και θα λειτουργεί χωρίς ρευστό και γι' αυτό οι καταναλωτές πρέπει να έχουν, ε, σε φυσικό χαρτονόμισμα δηλαδή, και γι' αυτό οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά η ενιαία αγορά συμπεριλαμβάνοντας όλους στο πεδίο το χρηματικό και το ε, χρηματοπιστωτικό. Σίγουρα οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Και σε αυτές τις χώρες θα έλεγα ότι το ίμιση ε, του πληθυσμού, του ενήλικου πληθυσμού, δεν έχει αυτή τη στιγμή ε, τραπεζικό λογαριασμό. 30 εκατομμύρια άνθρωποι ενήλικοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό και 6-7 εκατομμύρια ενήλικες έχουν κάνει αίτηση ανοίγματο τραπεζικού λογαριασμού και ε, δέχθηκαν αρνητική απάντηση απάντηση. Προφανώς ε, όσοι έχουν πληγεί, έχουν χαμηλά εισοδήματα ή εισοδήματα που προκύπτουν σε μη τακτά χρονικά διαστήματα ή είχαν προκύψει προβλήματα στην ε, παρελθούσα πορεία τους. Βεβαίως είναι ανεπαρκείς, ανεπαρκείς οι υποδομές τραπεζικής και πληρωμών σε ορισμένες χώρες μέλη. Μπορεί να μην έχουν επαρκή πληροφόρηση ή μόρφωση οι, ετούντος, ετούντες, αλλά και μπορεί να μην έχουν και αυτή την συνήθεια. Ε, όλοι, όλες αυτές είναι οι αιτίες. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη, εποχιακοί ε, εργαζόμενοι σε τακτικές, αυτή χρονική βάση φοιτητέ, μεταξύ άλλων, έχουν υποβάλει διάφορα παράπονα κατά καιρού. Και εγώ έχω προσωπική εμπειρία. Ε, είχα τεράστιες ε, δυσκολίες να είχα ακούσει από έναν άνθρωπο του περιβάλλοντος μου, του πολύ στενού περιβάλλοντος μου, ο οποίος ε, πήγε στη χώρα προέλευσής του για να ε, σπουδάσει και δεν μπορούσε να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό γιατί θεωρείται ότι ερχόταν από το εξωτερικό στο πλαίσιο των σπουδών του. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές ότι η ενιαία αγορά δεν λειτουργεί για όλου. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά παραδείγματα δυσλειτουργιών. Και Σίγουρα οι τράπεζες χωρίζουν τους πελάτες σε εμπορικώς ελκυστικούς και εμπορικώς ε, μη ελκυστικούς. Οι πολίτες δυσκολεύονται εξαιρετικά να ανοίγουν και να λειτουργούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε άλλα κράτη-μέλη παρά την προφανή ευκολία του διαδικτύου. Έχουν την ε, δυνατότητα να κινούνται παντού στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια χάρη στις συνθήκες και σε όλη αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει εμείς και τελικά όταν ταξιδεύουν και κινούνται δυσκολεύονται πάρα πολύ να οργανώσουν την καθημερινότητά τους. Οι συνθήκες επιλεξιμότητας είναι πάρα πολύ περίπλοκες Ωστόσο, πολλά από αυτά τα προβλήματα προκαλούνται από νομοθετικά και κανονιστικά εμπόδια. Αυτά ε, ισχύουν, ο νόμος ισχύει. Ωστόσο, πολλά εμπόδια ε, οφείλονται σε επιχειρηματικές πρακτικές οι οποίες ε, βολεύουν μόνο την τράπεζα και οι οποίες έχουν να κάνουν με την προσδοκόμενη κερδοφορία ή την αξιολόγηση κινδύνου. Ξέρω ότι απογοητεύσαμε κάποια από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την έκδοση της αντί τη σύνταξη μιας νομοθετικής πρότασης εξ αρχής. Ωστόσο, πράγματι συμφωνούμε, χρειάζεται ένα άκαμπτο πλαίσιο ε, για τα ε, πρότυπα σύγκλησης ώστε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες. Κάποια κρατημέλη έχουν νομοθετήσει για το θέμα αυτό. Κάποια άλλα κρατημέλη έχουν αφήσει ε, τον κλάδο να το ρυθμίσει ε, θεσπίζοντας ορισμένους κανόνες ε, δεοντολογίας και ερχόμενα σε συμφωνία με τον εκάστοτε τραπεζικό κλάδο. Σε άλλα κρατημέλη δεν έχει γίνει κανένα απολύτω βήμα. Αυτά τα γνωρίζετε. Όπως γνωρίζετε, εμείς εκδώσαμε μία σύσταση στην οποία λέγαμε ξεκάθαρα ότι αυτή η σύσταση είναι μόνο ένα πρώτο βήμα και αν τελικά αποδειχθεί ότι η σύσταση αυτή δεν έχει την ευεργετική επίδραση την οποία εμείς επιθυμούμε, τότε θα αντλήσουμε τα διδάγματα από αυτή την αποτυχία. Με άλλα λόγια, ότι δηλαδή θα προτείνουμε την υιοθέτηση νομοθετικής πράξης. Και ελπίζουμε ότι η σύσταση αυτή έχει στείλει ένα σαφές μήνυμα στα κράτη-μέλη και στον τραπεζικό κόσμο, ότι δηλαδή αυτή η δυσλειτουργία, η έλλειψη ε, της αγοράς πρέπει να ε, σταματήσει πλέον να υπάρχει και θα πρέπει το, η πρόσβαση στην τραπεζική να είναι δικαίωμα το οποίο να παρέχεται σε όλους. Στη σύσταση προτείνουμε τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος σε τοπικό επίπεδο για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων. Ωστόσο, με πολύ ε, σταθερό και επίμονο τρόπο αναφερόμαστε στις συνθήκες και στις προϋποθέσεις. Δεν θα πρέπει ας πούμε, η πρόσβαση σε λογαριασμό να ε, ε, ε τη χάνει άρνησης για λόγους ε, για λόγους καθεστώτος απασχόλησης μεταξύ άλλων. Και λέμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει το ζήτημα τον Ιούλιο του 2012 τα κράτη-μέλη υποβάλλουν αναφορές για το κατά πόσο συμμορφούνται ή όχι με την λόγω σύσταση και περιμένουμε ότι η τελική έκθεση θα συνταχθεί αυτόν τον ε, μήνα. Θα αναλύσουμε τότε τι θα έχει αλλάξει και τι ενδεχομένως δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Αυτό πολύ φοβούμε ότι θα είναι η αλήθεια για ορισμένα κράτη-μέλη και μετά θα επανεξετάσουμε τη θέση μας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί ε, με τα συνοδά μέτρα. Το καλοκαίρι αυτά. Επομένως, με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη δουλειά σας να σας πω ότι υπάρχουν διάφορα άλλα ζητήματα λιανικής τραπεζικής τα οποία εξετάζουμε. Για παράδειγμα, η διαφάνεια ως προς, τις, ε, ε, ως προς τα τέλη και τα έξοδα ε, την ε, αλλαγή του κόστους και την αντιστροφή, όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος της δέσμης χρηματοπιστωτικών μέτρων, η οποία ως πρόταση, πρόταση θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν βεβαίως από την πρόοδο που θα έχουν σημειώσει κατά την άποψή μας τα κράτη-μέλη, ε, προσπαθώντας να συμμορφωθούν με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε αποφασισμένοι να δράσουμε και βεβαίως από την άλλη ε, θα πάρουμε όλο το χρόνο που θα χρειαστεί για να εξετάσουμε τα δεδομένα, τα στοιχεία και τελικά να καταλήξουμε μήπως είναι η νομοθεσία η καλύτερη άγουσα. Ε, προς το παρόν εμένουμε στη σύσταση, μπορεί όμως να χρειαστεί νομοθεσία. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα και ε, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας για την ευκαιρία που μας δίνεται να παραστούμε σε αυτή την ακρόαση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ξεκάθαρες δηλώσεις σας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζουμε και εμείς να ε, τροφοδοτήσουμε τη δουλειά σας με τα δικά μας ε, στοιχεία. Να προχωρήσουμε λοιπόν στην πρώτη συνεδρία, σε αυτή την ακρόαση. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να μπορώ να καλωσορίζω τους διακεκριμένους εμπειρογνώμονές μας. Θα μιλήσουμε για τη βασική τραπεζική ως ε, δικαίωμα του καταναλωτή και ως καθολική υπηρεσία, ωφέλη και ε, από την ε, χρηματοδοτική συμπερίληψη αν θέλετε και μειονεκτήματα λόγω του τραπεζικού αποκλεισμού. Θα ακούσουμε ε, λοιπόν την κυρία Αν Φάιλε, επικεφαλής του Τμήματος Νομικών και Οικονομικών Υποθέσεων του BUC, e BEUC, που είναι η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών. Θα ακούσουμε τον κύριο Ούντο Ράιφνερ, καθηγητή εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και ε, διευθυντή του τμήματος έρευνας ε, του ανεξάρτητου αυτού ε, Ιδρύματος για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες. Θα ακούσουμε τον κύριο Βίκτορ Καμίνσκι, αντιπρόεδρο της Εθνικής Ένωσης των Συνεταιριστικών Οργανισμών για τις Αποταμιεύσεις, των Συνεταιριστικών Αποταμιευτικών Τραπεζών δηλαδή και των Ενώσεων Οργανισμών Χορήγησης Πιστώσεων από το Σόποτ της Πολωνίας και τον κύριο Πίτ Πίτερ από τη Δανία που ε, είναι στέλεχος στην Advocat Firmet Shots AS, νομικό ε, ε, σύμβουλο σε δικηγορική εταιρεία, ο οποίος θα μας εκθέσει την νομική σκοπιά της υπόθεσης. Θα έχουμε σχόλια και θα μπορέσετε εσείς να απαντήσετε, αλλά και βεβαίως να σχολιάσετε και τις τοποθετήσεις των άλλων. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Αν Φάιλι. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου έχετε απευθύνει να παραστώ σε αυτή την ακρόαση. Θα επαναλάβω κάποια πράγματα τα οποία έχουν ήδη λεχθεί, αλλά με τα οποία συμφωνούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 30 εκατομμύρια άτομα άνω των 18 ετών δεν έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο ε, λογαριασμό. Βεβαίω είναι ένα πρόβλημα που αφορά πολύ περισσότερο ορισμένα κράτη-μέλη παρά άλλα, αλλά αφορά και χώρες που η τραπεζική είναι σε αρκετά προηγμένα επίπεδα. Στη Γαλλία ε, 750.000 Γάλλοι δεν έχουν δικαίωμα να έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό αυτό τη στιγμή και αυτό το νούμερο είναι αρκετά υψηλό. Σίγουρα το σύστημα σε αυτή τη χώρα είναι πολύ περίπλοκο, είναι λίγο γνωστό και δεν αξιοποιείται. Δηλαδή δεν προσφεύγουν ενώ το δικαιούνται ε, πάρα πολλοί άνθρωποι και τελικά προσφεύγουν λιγότερο, λιγότεροι από 30.000 άνθρωποι το χρόνο ενώ θα μπορούσαν κατά της αρνητικής απόφασης αυτής. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που ποτέ δεν είχαν τραπεζικό λογαριασμό, αλλά και άνθρωποι που είχαν και τελικά τους αρνούνται οι τράπεζες κάποια στιγμή χρονική και μετά δεν μπορούν ποτέ ξανά να έχουν ε, τραπεζικό λογαριασμό. Η ύπαρξη όμως ε, τρεχούμενου λογαριασμού είναι απαραίτητη έτσι ώστε ε, να, ενσωματώνονται όλοι στην κοινωνία στην οποία ζουν. Ο κοινωνικός αποκλεισμός πηγαίνει χέρι-χέρι με τον χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό. Δεν μπορεί κανείς πρόσβαση στην πίστοση, στην ασφάλιση, ε, σε αποταμιευτικά προϊόντα. Άλλωστε, οι μετανάστες εργαζόμενοι που θέλουν να αποστείλουν χρήματα στις οικογένειές τους μπορούν να στείλουν χρήματα μόνο της Western Union, για παράδειγμα, και τέτοιων σχετικών ε, επιχειρήσεων, οι οποίες όμως χρεώνουν πάρα πολύ ψηλά τα εμβάσματα αυτά, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μισθούς, σε συντάξεις, σε ε, παροχή κοινωνικής ασφάλισης. Δεν είναι δυνατόν ε, να πληρώσει κανείς σε ρευστό, σε φυσικό χρήμα, φυσικό χαρτονόμισμα. Πολύ δύσκολο μπορεί κανείς να πληρώσει το νίκη του ε, μόνο με χαρτονομίσματα. Περιπλέκεται η πληρωμή των λογαριασμών. Να πληρώσει κανείς με χαρτονομίσματα, να περιμένει τόσο πολύ ώρα για να πληρώσει με χαρτονομίσματα το λογαριασμό του νερού, ε, του ρεύματος, του τηλέφωνου, είναι κάτι που δυσχεραίνει τη ζωή του. Και βεβαίως δεν μπορεί να υποφεληθεί από τις πωλήσει στο διαδίκτυο, διότι η κάρτα πληρωμών πιστοτική ή χρεωστική παραμένει το βασικό μέσο πληρωμής στο διαδίκτυο. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα όσοι εργάζονται σε άλλα κράτη-μέλη βλέπουν τη ζωή τους να περιπλέκεται πάρα πολύ αν δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Ο κύριος Τζόναθαν Φόλ ε, παρουσίασε το παράδειγμα μέλους του περιβάλλοντο του, του στενού και εγώ έχω το ίδιο παράδειγμα να πω. Ε, στην Σουηδία δεν μπόρεσε ε, να ανοίξει η κόρη φίλης μας λογαριασμό γιατί θα έμενε κάτω από δύο χρόνια. Και πρέπει να ε, κάνει ανάληψη από ATM για να κάνει οποιαδήποτε πληρωμή. Δηλαδή κάθε φορά που κάνει ε, ανάληψη από ATM του παίρνουν προμήθεια και βεβαίως έχει πάρα πολύ υψηλό ετήσιο κόστος με όλες αυτές τις αναλήψεις ε, που πρέπει να κάνει για να κάνει τις καθημερινές του ε, πληρωμές. Ακριβώς γιατί δεν μπορεί να έχει τραπεζικό λογαριασμό στη χώρα αυτή και πρέπει να κάνει αναλήψεις από το ETM, από τον λογαριασμό της χώρας από την οποία προέρχεται. Βεβαίως ε, συνεχώς μιλούμε για τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλες ε, χώρες μέλη, όμως είναι αδύνατη η αποστολή του να ανοίξει κανείς λογαριασμό σε μια άλλη χώρα, ε, πόσο μάλλον όταν δεν είναι κάτοικος ε, της χώρας αυτής. Και αν δούμε τη, χρεώσεις των τραπεζών βλέπουμε ότι ο καταναλωτής θα μπορούσε να επωφεληθεί εξαιρετικά από το να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό σε γειτονική χώρα και κυρίως μέσω διαδικτύου. Μιλούμε για έναν κατακαιρματισμό της ενιαίας αγοράς ω ε, ως προς τον ε, κλάδο της τραπεζικής θα μπορεί και θα πρέπει ο καταναλωτής να καταθέτει και να αποσύρει χρήματα, να κάνει πληρωμές, να εκτελεί και να δίνει εντολές πληρωμής για να πληρώσει τους λογαριασμούς του, να κάνει εμβάσματα σε τρίτους ε, ή να δίνει αυτόματη εντολή χρέωσης του λογαριασμού του, να κάνει αγορές να έχει πρόσβαση στα ATM για να κάνει αναλήψεις και για να κάνει πληρωμές και θα πρέπει να λαμβάνει τα statements σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μπορεί να παρακολουθεί τις συναλλαγές του και θα πρέπει να του προσφέρεται αυτή η κίνηση λογαριασμού και σε διαδικτυακό επίπεδο. Και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνήθειες που ε, επικρατούν σε κάποια χώρα, δηλαδή να προσθεθούν ε, επιπρόσθετες ε, δυνατότητες και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ορισμένες χώρες έχουν προβλέψει τη δυνατότητα υπερανάληψης, κάτι το οποίο εγώ απέφχομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υφίσταται σε πολύ συγκεκριμένο και προκαθορισμένο πλαίσιο. Και ενδεχομένως όλα αυτά θα πρέπει να προσφέρονται δωρεάν σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων. Και για να μην Ε, υπάρχει στίγμα στα άτομα, θα πρέπει ένας πάροχος να προσφέρει όλες αυτές τις υπηρεσίες που θα πρέπει να ε, είναι συνδεδεμένες με ένα βασικό λογαριασμό, τραπεζικό λογαριασμό. Ε, οργάνωση την οποία εκπροσωπώ εκφράζει τη λύπη της γιατί η Επιτροπή δεν πρότεινε ένα δεσμευτικό νομοθετικό κείμενο. Πρότεινε το soft law, δηλαδή μια σύσταση μη υποχρεωτικού χαρακτήρα, κάτι το οποίο δεν λειτουργεί κατά την άποψή μας. Θα παρακολουθήσουμε εκ του σύναγκης το κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα συμμορφωθούν με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από εκεί και πέρα θα ήθελα ε, να κάνω ένα παραλληλισμό με το δικαίωμα πρόσβαση στο διαδίκτυο, το οποίο θεωρείται θεμελιώδες ε, δικαίωμα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει ενδεχομένως να αναγνωριστεί το δικαίωμα πρόσβασης σε ένα τραπεζικό ε, λογαριασμό ως θεμελιώδες ε, δικαίωμα των ανθρώπων. Μπορεί κανείς να ζήσει και χωρίς διαδίκτυο, όχι καλά, αλλά να ζήσει, εν πάση περιπτώσει. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τραπεζικό λογαριασμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και ένα αντίγραφο της έκθεσης να σας δώσουμε, ώστε να το έχετε στο υπόλοιπο συνέχεια τη συζήτηση. Καθηγητή Ράιφνα, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Δουλεύω πάνω σε αυτό το θέμα είχα ξεκινήσει τη δεκαετία του 80 στις είπα ότι μιλούσαμε για banking, τραπεζικές λογαριασμούς διαμέσεις της, καθ' όλη διάρκεια ζωής και υπάρχουν ακόμα αποφάσεις που δεν πέρασαν στο νότο δικαστήριο μετά στην διάρκεια της Φιλανδικής και της Βελγικής ε, Προεδρίας έρχεται ένας αρχικός προβληματισμός για βασική πρόβλημα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τελικά ούτε και τότε πέρασε. Είχαμε ένα διεθνές συνέδριο με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης 5 στο Γκέτεμπουργκ, πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συζητήσαμε τα θέματα και μετά στη Γερμανία έγινε μια ευρία δημόσια συζήτηση που τελικά οδήγησε στην ε, εν λόγω σύσταση. Και εδώ τρία χρόνια έχουμε αξιολόγηση. Και τελευταία ήταν αρνητική αξιολόγηση κατά από την κυβέρνηση. Το ερώτημα λοιπόν είναι <laughs> εξαιρετικά πιο πολύπλοκο από ό,τι εμφανίζεται εδώ. Το να έχει κανείς ή να μην έχει τραπεζικό λογαριασμό δεν, δεν υποδηλεί τίποτα απολύτως. Γιατί με αυτού του είδους τα εμπειρικά στοιχεία που έχουμε εδώ πέρα εδώ, για παράδειγμα, ερώτημα που υπάρχει, το βρίσκεται δύσκολο να, έχει, να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό. Εάν κάποιος έχει ήδη δύο και θέλει να πετύχει ένα τρίτο, θα απαντήσει ναι. Ναι, το βρίσκω δύσκολο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η τράπεζα θα έλεγε πρέπει να είναι δύσκολο, δεν μπορούμε να βγάλουμε χρήματα με, ε, με τρεις λογαριασμούς. Και εγώ είμαι ένα θύμα αυτό. Δεν είναι ο πρωτογόνη. Θα σα κάνουμε να, να, να πληρώσετε για του υπόλοιπου λογαριασμού που δεν είναι ο βασικό τροφοδότη λογαριασμό, σα μου είπαν. Έκανα λοιπόν μια μελέτη και λόγω παρανόηση δεν έχει, την έχετε λάβει ακόμα, όπου όλα τα επιχειρήματα που ακούστηκαν υπάρχουν εκεί πέρα και είναι μια σύνοψη των συζητήσεων και των ερευνών. Απολύτει από τρία κομμάτια εργασία αυτή. Το ένα κομμάτι είναι οι πολιτικές επιλογές. Όχι, δεν μπορείτε να διαβάσετε. Οι πολιτικές επιλογές. Το δεύτερο είναι πού θα πρέπει να βασίζεται στην χρηματοοικονομική κρίση και τις αρνητικές διακρίσεις. Και το τρίτο κομμάτι, ποιες είναι οι λύσεις, ποιες είναι οι επιλογές. Ξεκινώ με τις πολιτικές επιλογές. Η έλλειψη, ε, έλλειψη πρόσβασης σε έναν τραπεζικό λογαριασμό για όλες τις συναλλαγές στην Ευρώπη ποικίλει από το 17% έως το 1%. Πολλοί όμως μπορούν να απαντήσουν ότι δεν το χρειάζονται θεωρούν ότι το κόστος είναι πολύ υψηλό. Τώρα στα θέματα περί αποκλεισμού δεν ξέρουμε γιατί ξαναγκάλυψε κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε περιοχές όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία όπου δεν υπάρχει καν τραπεζικό υποκατάστημα και έχουμε επομένω άτομα που δεν είναι στεδεμένα με τις τράπεζες που αυτό συμβαίνει σε υποαναπτυκτές χώρε αλλά και σε εξαιρετικά ανεπτυγμένε όπως στην Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο που υπάρχουν πάρα πολλέ τράπεζε και υποκαταστήματα οπότε που όμως εκεί υποκρίνουν ότι δεν είναι αρκετά ε, κερδοφόροι οι πελάτες τους, κάποια στρώματα δηλαδή, τους αποκλείουν. Μπορούμε να βρούμε κάποια σχετικά στοιχεία. Διαβάστε το. Έχετε εδώ πέρα την σχέση μεταξύ της κοινωνικής τάξης και της ε, ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού. Αυτή είναι η υπομελέτη στον του 2010. Βλέπετε ότι αυτοί που έχουν υψηλό εισόδημα έχουν ε, η αναλογία αυτών που έχουν ε, τραπεζικό λογαριασμό είναι 10 προς 1 σε σχέση με τους φτωχούς. Είναι δηλαδή οικονομικό πρόβλημα, ταυτόχρονα και κοινωνικό. Απ' την άλλη όμως η ίδια η κοινωνία χρειάζεται και θέλει τους ανθρώπους να έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Όταν κάναμε αυτή τη συζήτηση στη Γερμανία, είχαμε κάποιε στατιστικές που μας απεκάλυψαν πόσα εκατομμύρια πρέπει να δαπανούν σε άτομα, γιατί θέλουν να του καταβάλουν ε, τα επιδόματα ανεργία ή άλλα ε, προνοιακά επιδόματα μετρητή, γιατί δεν είχαν ε, τραπεζικό λογαριασμό. Και αυτό του τύχησε πολλά εκατομμύρια. Είναι πολύ πιο φθηνό, ιδιαίτερα με την αυτόματη καταβολή πληρωμών ή προνοιακών επιδομάτων, είναι πολύ πιο φθηνό εάν υπάρχει τραπεζικό λογαριασμό. Ένα άλλο θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ψωμιού και βουτυριού στην τράπεζα. Δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη ε, για τραπεζικό λογαριασμό όσο χρειάζεσαι να έχεις ε, ηλεκτρισμό και νερό. Είναι εργαλείο ο τραπεζικός και το πόσο χρησιμοποιείται το εργαλείο αυτό εξαρτάται το περιβάλλον και τις ανάγκες και τις συνθήκες του άτομα. Χρειαζόμαστε λοιπόν εμπειρικά να δούμε πού βρίσκονται τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε όμως με τα υφιστάμενα εμπειρικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει. Τα περισσότερα έχουν προκύψει από δημοσκοπήσεις ιδιαίτερα της Eurostat. Δεν νομίζω όμως ότι οι κοινωνικές έρευνες μπορούν να γίνονται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό άπτεται του marketing, όχι της κοινωνικής έρευνας. Εάν ρωτάς κάποιον αισθάνεστε καλά ή κακά, δεν μπορεί να μας αποδώσει και να μας πει σωστά απαραίτητα το τι υπάρχει. Ως κοινωνιολόγος που έχω δει πάρα πολλά εμπειρικά στοιχεία, βλέπω αυτή την παράξενη τάση να ρωτούν τη γνώμη των ανθρώπων. Ενώ το απτό στοιχείο είναι ποιοι έχουν πεζικό λογαριασμό και μετά να δούμε ποιο είναι ο λόγο που δεν έχουν. Οπότε μετά μπορούμε να εντοπίσουμε αν υπάρχει πραγματικά το πρόβλημα ή όχι. Ω λύση βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν οι άνθρωποι δεν το βρίσκουν ε, σωστό, το βρίσκουν ε, αν θέλετε δεν, δεν τους διευκολύνει, ας τους διδάξουμε. Εάν οι άνθρωποι το βρίσκουν πολύ δαπανηρό το να έχουν τραπεζικό λογαριασμό, ότι πρέπει να το περικόψουμε το κόστο. Άνθρωποι μπορεί να μην έχουν πρόσβαση γιατί είναι υπερχρεωμένοι. Οπότε πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Η πρότασή μου, εδώ και 30 χρόνια είναι η ίδια, ότι πρέπει να εστιάσουμε στο πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι η υπερχρέωση. Το υπερχρέωση είναι κοινωνικό πρόβλημα του να μην έχει τραπεζικό λογαριασμό και τίποτα άλλο. Το ΕΛΚ έχει μια παράδοση του 2004 που όπως ξέρετε τότε ήταν η χρονιά όπου το ΕΛΚ άλλαξε την οδηγία, ε, το προσχέδιο της οδηγίας του 2004 και ο στόχος ήταν η εξάλληψη της υπερχρέωσης. Και με τη νέα οδηγία είχαμε και την ε, οδηγία ε, του εξαιρετικά υψηλού ε, το κοφόρο λογαριασμού όταν ε, έχει εκπνεύσει προθεσμία ε, καταβολής και εξόφλησης του, της υπερχρέωσής σας. Το θέμα λοιπόν πραγματικά είναι τι πρέπει να κάνουμε ώστε τα αποτελέσματα της υπερχρέωσης να μην εμποδίζουν και να επιδεινώνουν την κατάσταση των ε, ανθρώπων στον τομέα της χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Γιατί τα πάντα συνδέονται με την ε, αξιοπιστία σου, την πιστοληπτική σου ικανότητα. Εάν χάσει την πιστοληπτική σου ικανότητα δεν σε καλός πελάτης. Από πού κάνουν τα χρήματά τους οι τράπεζες. Ο τραπεζικό λογαριασμό, αν θέλετε, είναι το κέντρο κερδοφορία για τι τράπεζε. Γιατί? Γιατί τυχαίνεις, παίρνεις ένα πελάτη, στον οποίο στη συνέχεια μπορούν να τους πωλήσει προϊόντα και ένας από τα πιο συχνά θέματα είναι η υπερχρέωση μέσω των χρεωστικών καρτών και όλα αυτά φέρνουν εισόδημα στους, στις τράπεζες. Βέβαια οι φτωχοί άνθρωποι δεν μπορούν να υπερχρεωθούν, ούτε και θα έπρεπε να του επιτρώξει, επομένω δεν μπορεί να κάνει χρήματα. Η αγορά λοιπόν είναι μια αστοχία τη αγορά. Δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα αυτό η αγορά. Και αυτό προκύπτει και η οδηγία, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν τραπεζικό λογαριασμό εκεί που τους συμφέρει. Εκεί που υπάρχει αστοχία της αγοράς χρειαζόμαστε συγκεκριμένες συστάσεις και ε, οδηγίες, συγγνώμη, και ε, νομοθεσία. Τι χρειάζονται αυτοί οι υπερχρεωμένοι άνθρωποι. Το ερώτημα είναι ποια είναι η λειτουργία του τραπεζικού λογαριασμού σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτούς τους ανθρώπους υπερχρεωμένους φαίνεται ότι μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες είναι να τηρείται η ρευστότητα και να τηρούνται τα οικονομικά του σπιτιού. Να ξέρεις πού είναι το έσοδό σου και οι δαπάνε σου. Σου απευθύνεται, σου αποστέλλεται μία, ε, ένας απολογισμός κάθε μέρα. Και αυτό είναι, είναι θεμελιώδες για τη χρηματοοικονομική κατάσταση να έχει συνολική επισκόπηση. Ένα άλλο σημείο είναι το διαβατήριο. Ο τραπεζικό λογαριασμό είναι σαν το διαβατήριό σου. Έχει να κάνει με την, με την αξιοπρέπειά σου, με την ε, δημόσια εικόνα σου. Στη ΣΥΠΑ ιδιαίτερα και συγκεκριμένα και, και, κυριολεκτικά μια πιστοτική κάρτα είναι διαβατήριο. Είναι τραπεζική ταυτότητα. Εάν δεν έχεις τραπεζική κάρτα, εάν δεν έχεις ε, πιστοτική κάρτα, είσαι πολίτης δευτέρας κατηγορίας. Είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λοιπόν. Βέβαια, έχουμε και τους μετανάστες που ήδη αναφέρθηκαν. Οι μετανάστες έχουν τεράστιο πρόβλημα. Εάν δείτε τις τιμές που χρεώνουν η Western Union και όλα αυτά τα μαγαζιά που χρεώνουν για την, με τη, για την μεταφορά την, ε, χρημάτων είναι πραγματικά εξωφρενικά ποσά. Δηλαδή αυτοί που είναι ήδη φτωχοί χάνουν πάρα πολλά ακριβώς γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε ένα τραπεζικό λογαριασμό όπου η προμήθεια είναι δοξο Θεός ε, κάπως πιο μικρή και υπάρχει και κάποιος έλεγχος αν θέλετε της χρέωσης. Εάν υπάρχει λοιπόν μια λύση η λύση θα πρέπει να είναι, να είναι νόμιμη. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε την κατάσταση της τράπεζας που ε, χορηγεί τον τραπεζικό λογαριασμό, γιατί υπάρχουν ευαλωτότητες και για την τράπεζα. Γιατί ως πιστωτές θα πρέπει επίσης να τους ε, κοιτάξουμε. Έχω επίσης κάνει κρεσί σε ό,τι αφορά τις ε, πιστώσεις χρειάζεται και το όριο υπερανάληψης. Εξού και η σύσταση, συμφωνώ με αυτήν, με την ε, πρόσθεση θα, του ότι θα πρέπει να διευκρινίζεται και το κόστος και η συνολική πίστη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και επίσης ευχαριστούμε που μας θυμίσατε την μακρά ιστορία Τη πρόταση αυτή που δεν τη γνωρίζαμε για να ειλικρινέως, γιατί είμαι σε αυτήν την Επιτροπή τρία χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ για τον πλούτο τη εμπειρία σα, ίσως να υπάρξει τώρα κάποια πρόεδρο. Οι πάντε τώρα έχουν αναχειράσει και την εισήγησή σα, οπότε μπορούν να τη μελετήσουν. Επόμενος ε, ομιλητή για 10 λεπτά θα είναι ο κ. Καμίνσκι. Καλησπέρα Ευχαριστώ που, που ε, προσκαλέσατε και, τις, ε, ε, και την Ένωση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων να συμμετάσχουν στην ακρόαση αυτή. Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για το πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό και να κάνω κάποια σχόλια και προτάσεις στο παιδί αυτό. Εντάχει, να σας πω ότι προσωπεύω το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, των Πιστοτικών Ιδρυμάτων. Είναι πολλές οι χώρες οι οποίες εκπροσωπούνται. Για εκείνους που ίσως να μην είναι πολύ εξοικειωμένοι με τα συνδικάτα, πιστωτικά συνδικάτα, να σας πω ότι είναι ε, συντεχνίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. συνεταιρισμοί χρηματοπιστωτικών ιδρωμάτων. Οι βασικές αρχές είναι ότι λειτουργούμε τοπικά, ε, καθορίζοντας ε, με κάποιους κοινούς δεσμούς, ε, δηλαδή με τη βάση κριτηρίων όπως γεωγραφική περιοχή, η απασχόληση σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή η εταιρεία ή η ύπαρξη μελών σε συγκεκριμένους οργανισμούς. Οι ενώσεις αυτές, πιστοτικές ενώσεις, δεν λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση. Είμαστε δηλαδή, λειτουργούμε τοπικά και εξυπηρετούμε μόνο τα μέλη μας τοπικά. Ως μη κερδοσκοπικά θεσμικά όργανα, οι πιστοτικές ενώσεις διανέμουν ε, κάθε πλεόνασμα στα μέλη τους μέσω ε, προσιτών δανείων, μερισμάτων και ενίσχυσης ε, του κεφαλαίου των μελών του. Οι ενώσεις αυτές οι πιστοτικές παρέχουν διάφορες ε, εξυπηρετήσεις αποταμίευσης και επεκτείνουν τα, τα, τα δάνεια στα μέλη τους, ιδιαίτερα για ε, οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. οι πιστοτικέ ενώσει διαφέρουν από τι τράπεζε. Εμεί είμαστε μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, αλλά επίση διαφέρουν και από του μη κυβερνητικού οργανισμού ή μικρο χρηματοπιστωτικού οργανισμούς, γιατί οι ενώσει μα είναι αυθύπαρκτε, αυτόνομε, βασίζονται στη δική του χρηματοδότηση, δεν έχουμε εξωτερικού επενδυτέ, ούτε χρειαζόμαστε οποιαδήποτε εξωτερική υποστήριξη, ούτε χρησιμοποιούμε ε, κρατικές επιδοτήσεις για την ε, δουλειά μας και τις δραστηριότητε που αναπτύσσουμε. Κάποιες πιστοτικές ενώσεις δεν προσφέρουν μόνο απλές τραπεζικού τύπου υπηρεσίες, αλλά και υπηρεσίες όπως ε, υπηρεσίες πληρωμών, λογαριασμών όψεως, χρεωστικές κάρτες, αυτόματα μηχανήματα ανάληψης και ορισμένες μάλιστα και χρηματοδότηση ε, στεγαστικής πίστης. Όπως τόνισα και προηγουμένως, ε, αυτές οι ενός πιστοτικές ε, μπορούν να είναι πολύ μικρά χρηματοοικονομικά θεσμικά όργανα, τα οποία λειτουργούν στις περισσότερες περιπτώσεις σε εθελοντική βάση, από εθελοντές. Μόνο τα διοικητικά συμβούλια ή τα εποπτικά συμβούλια ε, αποτελούνται από άτομα τα οποία δεν έχουν λάβει καμία αμοιβή για δραστηριότητά τους. Οι πιστοτικές ενώσεις ε, ιδρύθηκαν για να παράσχουν στις ε, τοπικές κοινότητες προσπέλαση στην χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αποφεύγοντας ακριβώς τους καταχρηστικές δανειστικές εναλλακτικές που υπάρχουν. Σήμερα, σήμερα οι πιστοτικές ε, ενώσεις εξακολουθούν ε, να εστιάζουν σε χαμηλότερους, χαμηλού εισοδήματος καταναλωτές και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα άτομα εκείνα τα οποία ε, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα στην χρηματοδότησή τους θα πω κάποια πράγματα στις κυριότητές μας για να υποστηρίσουμε ακριβώς την πρωτοβουλία χρηματοοικονομικής ένταξης και ολοκλήρωσης. Θα ήθελα να πω λοιπόν σε σχέση με την λόγο πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αυτό που συστώνουμε είναι μια ολιστική προσέγγιση η οποία απαιτείται για να ενισχυθεί η χρηματοοικονομική αυτή ένταξη των πάντων. Και με ολιστική προσέγγιση εννοούμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, να είναι πληροφορημένοι, να τους παράσχουμε ε, συμβουλές ε, ό,τι αφορά την πρόσβαση σε διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όχι μόνο ενό τραπεζικού λογαριασμού και χρειάζονται και νομικά και τεχνικά όρια σε κάποια κράτη-μέλη και χρειαζόμαστε και πολύ καλά δάνεια, ε, δηλαδή με προσιτούς όρους που δεν θα καταλήγουν στην υπερχρέωση των καταναλωτών, ιδιαίτερα σε σχέση και με σύγκριση με τις εμπορικές τράπεζες που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό σε πάρα πολλές χώρες όπου υπάρχουν και δραστηριοποιούνται οι πιστοτικές ενώσεις. Αντιμετωπίζουμε επίσης τεχνικά και νομικά εμπόδια σε κάποια κράτη-μέλη που περιορίζουν την ικανότητα των πιστοτικών ενώσεων να παράσχουν πλήρες υπηρεσίες στους λογαριασμούς, ε, λογαριασμούς ε, των, των ε, πελατών. Οι πιστοτικές όμως ενώσεις σε κάποιες, αλλά όχι όλες ε, τις χώρες μέλη, προσφέρουν πλήρες υπηρεσίες χωρίς να χρεώνουν καμία αμοιβή ή προμήθεια με απόλυτα διαφανείς όρους, χωρίς να εφαρμόζουν ρήτρες ε, κυρώσεων κλπ. Δεν ε, προσφέρουμε βέβαια την δυνατότητα ε, υπερανάληψης, αλλά κάθε μέλος της Πιστοτικής Ένωσης μπορεί να κάνει αίτηση για να ζητήσει εκτεταμένες υπηρεσίες έχουν πρόσβαση, οπότε έχουν πρόσβαση όχι μόνο στις βασικές υπηρεσίες, αλλά αν το επιθυμούν, υπό συγκεκριμένους όλους και συνθήκες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πιο πολύπλοκες και ε, σε πιο πολύπλοκες ε, υπηρεσίες. Σε κάποιες χώρες όπως η Εστονία, η Ιρλανδία, η Ρουμανία, οι πιστοντικές ενώσεις έχουν κάποιους περιορισμούς στο, στην προσφορά τους σε τραχόμενους λογαριασμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις όπως η Εστονία και τη Ρουμανία οι πιστοτικές ενώσεις δεν έχουν εξιοδότηση να αποδέχονται τις λεγόμενες καταθέσεις των ε, πολιτών, ακόμα και των μελών τους. Σε άλλες περιπτώσεις, ο εθνικός νόμος περιορίζει τη δυνατότητα των μελών να αποσύρουν, να, κάνουν ανάληψη των κονδυλίων τους, εάν έχουν ε, ε, πάγιες και κρεμείς δανειακές υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει στην Ιρλανδία. Και επίσης η πρόσβαση σε υποδομή πληρωμής πολύ συχνά είναι εξαιρετικά δαπανηρή για τις πιστοτικές ενώσεις. Στην περίπτωση της Πολωνίας είδαμε ότι 23% του ενήλικα πληθυσμού στην Πολωνία δεν έχει τραπεζικούς λογαριασμούς για δύο κυρίως λόγους. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε ό,τι αφορά το υψηλό κόστος διατήρησης τραπεζικού λογαριασμού και η έλλειψη εμπιστοσύνη απέναντι στις τράπεζες. Όμως, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας, βρήκαμε επίσης ότι 54% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι απλώς δεν χρειάζονται λογαριασμό γιατί προτιμούν να λειτουργούν με χρήματα μετρητά. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό επίσης ατόμων, ερωτηθέντων, που εξέφρασαν την προσήμισή τους ή που είπαν ότι έχουν πολύ μικρό εισόδημα, δεν έχουν ε, αποταμιεύσεις, δεν έχουν τακτική καταβολή μισθών ή ότι το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό, πολύ υψηλότερο το κόστος από το όφελος και υπάρχει απειροελάχιστο ενδιαφέρον για αποταμίευση. Μόνο 2,6% των ερωτηθέντων απάντησε ότι αντιμετώπισαν άρνηση από τις τράπεζες να τους ανοίξει λογαριασμό λόγω έλλειψης μόνιμης θέσης εργασίας. Κάποιοι είπαν ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκες ε, οι υπηρεσίες των τραπεζών, αλλά δεν είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό. αφήνω άλλες δραστηριότητε των ενώσεών μας που είχαμε τα δύο τελευταία χρόνια. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζουμε τη διατήρηση και την άσκηση πίεση στα κράτη-μέλη προκειμένου να προαχθεί η συμπερίληψη όλων στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Συμφωνούμε και κάνουμε γενική έκκληση ότι οι συγκεκριμένες ε, ε, να μην είναι πάρα πολύ περιοριστικές, ώστε το συνολικό κόστος για την, ε, να μπορεί να είναι ε, προσιτό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια κοινή προσέγγιση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένου και το πρόβλημά των υπερχρέωσης, δουλεύοντα με τρόπο που θα αντιμετωπίζεται υπερβολικό κόστος. Ο κανόνας κατά του ξεπλήματος ε, χρήματος δεν θα πρέπει να θέτει απαιτήσει που ίσως καθιστούν εμπόδιο ε, και μη προσέγγιση των ε, πιστοτικών ενώσεων σε σχέση με την μη ύπαρξη υποδομή είναι επίση ένα εμπόδιο για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Σε ορισμένε περιπτώσει, τεχνική βοήθεια μπορεί να υπάρξει είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από την εθνική κυβέρνηση κράτου ομιλή, ώστε να επεκτείνει τη λειτουργία τη δραστηριότητά τη τέτοιου είδου χρηματοπιστωτική ένωση. Ευχαριστώ πολύ που μας, για την εμπειρογνωμοσύνη στο πεδίο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ και ο καθηγητής Ράιφνερ αναφέρθηκε σε θέματα της ε, οδηγίας ε, περιπίστης. Η Επιτροπή αυτή έχει δεσμευθεί ακριβώς να αναθεωρήσει την οδηγία αυτή αυτή τη στιγμή και είχα μια σχετική παρουσίαση και μελέτη του θέματος χθες. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια σημεία που επικαλύπτονται και θα ζητήσουμε και από τον εισήγητη να μελετήσει. Και τελική παρουσίαση στη συνεδρία αυτή είναι από τον κύριο Πίτερ Ντιέρμπερκ. Ελπίζω να, να αναφέρω σωστά το όνομά σας. Να μας δώσετε και εσείς την πολύτιμη εμπειρία σας πάνω στο θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Εν συντομία θα αναφερθώ στις διατάξεις της συνθήκης, οι οποίες είναι σχετικές ε, με την προσπάθεια ρύθμισης της ε, πρόσβασης ε, σε τραπεζικό λογαριασμό ως ένα πεδίο γενικού οικονομικού συμφέροντος. Θα δούμε τα άρθρα, θα εξετάσουμε τα προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν και θα προσπαθήσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα. Έχω κάποιες διαφάνειες να σας δείξω Not on the screen. No. Oh, okay. Καλώς. Υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα και δεν προβάλλονται διαφάνειες στην οθόνη. Θα τα καταφέρουμε και χωρίς αυτές. Η πρώτη διάταξη που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι μια διάταξη που υπήρχε στην αρχική συνθήκη στο τμήμα περί κανόνων ανταγωνισμού. Μιλούμε για το άρθρο 106 της συνθήκης της ε, ε, υφιστάμενης συνθήκης σε σχέση με, τις, ε, ε, με τους φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Είναι εφαρμόσιμοι οι κανόνες, οι κανονικοί κανόνες που προβλέπονται από τη συνθήκη σε υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το γενικό οικονομικό συμφέρον ή ενδιαφέρον. Εάν θέλει κανείς να φύγει από αυτό το πεδίο εφαρμογής, τότε θα πρέπει να το τεκμηριώσει και να αποδείξει ότι δεν κάνει δυσανάλογη ε, παρίσφρηση ε, στους ε, κανονικούς κανόνες της ηθίκης, οι οποίοι είναι, επαναλαμβάνω, η ελεύθερη κυκλοφορία και ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, το SGI, ε, General Economic Interest, Γενικό Οικονομικό Συμφέρον, θεωρήθηκε εξαίρεση η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται. Και μετά πάμε στην ε, διάταξη που έχει να κάνει με τις υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος. Είναι μια διάταξη ε, την οποία εξέτασε περαιτέρω και ανέπτυξε η συνθήκη της Λισαβόνας. Στη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε το άρθρο 14 και είναι κρίμα που δεν μπορούμε να το προβάλλουμε στην οθόνη γιατί ήταν ένα από τα γλωσσικά αριστουργήματα της ε, συνθήκης ε, στα οποία, ε, τα οποία εμείς πράγματι μπορούμε να δημιουργήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέτοιου είδους γλωσσικά αριστουργήματα αριστούργήματα. Προκαλεί πονοκέφαλο και μόνο η ανάγνωση του άρθρου αυτού. Δεν είμαι σίγουρος ότι το αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει κάποιος που να το καταλαβαίνει πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει λέει αυτό το άρθρο ότι η Ένωση μπορεί να θεσπίσει τις αρχές για την λειτουργία των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή θα παράσχουν και θα χρηματοδοτήσουν αντιστοίχους τέτοιου είδους υπηρεσίες και μετά έχουμε ένα σωρό επιφυλάξεις ε, ε, ε, και το καθεξής. Όμως η αρχή είναι αυτή που σας ανέφερα. Ορισμένοι θα παρατηρήσετε ότι το άρθρο λέει ότι δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργεί υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Επομένως, σίγουρα θα προκύψουν διάφοροι δικηγόροι στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, οι οποίοι θα γύρουν εμφιβολίες κατά πόσο μπορεί κανείς να βασιστεί σε αυτό το άρθρο νομικός, ούτω ώστε να δημιουργήσει υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Και αξίζει να σημειώσουμε κάτι στο άρθρο 14, ότι δηλαδή το μέσο ρύθμισης αυτού του πεδίου πρέπει να είναι ένας κανονισμός. Σήμερα ακούσαμε εδώ να γίνεται αναφορά στο κανονιστικό πεδίο το οποίο είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και το οποίο διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη. Και έτσι λογικό είναι να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ε, το νομοθέτημα για τη ρύθμιση αυτού του θέματος είναι μία οδηγία, διότι η οδηγία λαμβάνει καλύτερα υπόψη της τις διαφορές στο νομικό πεδίο που έχει το κάθε από τα 27 κράτη-μέλη. Επομένως, εάν ήθελε κάποιος να χρησιμοποιήσει το άρθρο 14 και να βασιστεί σε αυτό, τότε θα προέκυπτε το εξής πρόβλημα, ότι το μόνο είδους νομοθέτημα που προβλέπεται είναι, μία, ένας κανονισμός. Λέει ο μιλητής. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να ε, βασίσει κανονισμό στο άρθρο 14. Και μετά έχουμε τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος στο πρωτόκολλο υπαριθμών 26 το οποίο πρωτόκολλο υπαριθμών 26 δεν μπορεί φυσικά να ε, συγκροτήσει νομική βάση για νομοθέτημα. Αξίζει όμως να αναφορθεί γιατί και εδώ για άλλη μια φορά έχουμε το ρόλο των εθνικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών οι οποίες έχουν ως ρόλο να παρέχουν, να αναθέσουν και να διοργανώσουν όλες αυτές τις ε, υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Δηλαδή η γλωσσική διατύπωση για άλλη μια φορά ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η δημιουργία ε, τέτοιου είδους υπηρεσιών. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι έχουμε τις υπηρεσίες γενικού ε, οικονομικού συμφέροντος στο ε, παράγωγο δίκαιο. Όταν ξεκινήσαμε με την απελευθέρωση της αγοράς, ε, οι βιομηχανίες που είχαν να κάνουν με το διαδίκτυο, με τις τηλεπικοινωνίες, με τη δικτύωση και γενικότερα με όλο αυτό το πεδίο, ε, στα νομοθετήματα του παράγωγου δικαίου είχαμε διατάξεις για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος πάντοτε. Υπάρχει δηλαδή νομολογία εκεί. Όμως να σημειώσουμε ότι σε αυτού του είδους τα νομοθετήματα δεν υπησέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι αυτή που δημιουργεί την υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος. Λέει η Ένωση ότι θα απελευθερώσουμε την εν λόγω αγορά και μετά θα θα σεβαστούμε τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος που θα θέλει να έχει το κράτος μέλος. Δηλαδή τηλεπικοινωνία σε απομακρυσμένες περιοχές, ε, τηλεφωνία σε απομακρυσμένες περιοχές και ούτω καθεξής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, σεβόμαστε ως Ένωση τις υπηρεσίες της εν λόγω που, δημιουργούν, που δημιουργούν τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η διατύπωση ε, στην ομολογία σε νομοθετήματα παράγωγου δικαίου. Δεν υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο προηγούμενο, νομικό προηγούμενο πάνω στο οποίο θα μπορούσαμε να εδράσουμε ε, τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος σε ε, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να δούμε επίσης το άρθρο 1.1.4 της διατάξης για την εναρμόνιση. Αυτό είναι το τελευταίο μας εργαλείο. Είναι και αυτό μια δυνατότητα, το άρθρο 114. Το κατά πόσο θα είναι χρήσιμο, αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα διατυπώσει κάποιος το τελικό μέσο το οποίο αποσκοπεί να υιοθετήσει. Θα θυμάστε ότι το 114 είναι μια διατάξη για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Επομένως, ως νομικός ε, θα προτιμούσα εγώ και διάφοροι άλλοι να έχουμε ξεκάθαρα την διασυνοριακή διάσταση παρούσα εκεί. Στο βαθμό που γίνεται πάρα πολύ μεγάλος λόγος για την κοινωνική συμπερίληψη, η οποία είναι ένας στόχος καθόλου σεβαστός, να μην παρεξηγηθώ. Καθόλου σεβαστός είναι αυτός ο στόχος. Ποια είναι όμως η διασυνοριακή διάσταση της κοινωνικής συμπερίληψης. Εάν τονίσει κανείς την πτυχή της κοινωνικής συμπερίληψης, της ενσωμάτωσης στην κοινωνία, τότε θα προσκρεούει σε εμπόδιο κάθε φορά που θα θέλει να ε, αξιοποιήσει το άρθρο 1114 ως νομική βάση. Θα ήταν καλύτερο να αξιοποιήσει το άρθρο 114 ως νομική βάση για να τονίσει ε, τις καταστάσεις ε, για τις οποίες μίλησαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι εμπειρογνώμονες, δηλαδή τη διασυνοριακή προβληματικότητα, όπως η κόρη της φίλης της εισηγήτριας της εμπειρογνώμονας που δεν μπορούσε να ανοίξει λογαριασμό στη Σουηδία ενώ θα έμενε εκεί, αν και όχι πάνω από δύο χρόνια, ή ο γιος του Τζόναθαν Φόλ, ο οποίος δυσκολεύτηκε να ανοίξει λογαριασμό όταν επέστρεψε στην πατρίδα του και το καθεξής. Ε, Αυτά θα τεκμηρίωναν τη χρήση του 114 ως νομικής βάσης. Αυτά είχα να σας πω για το νομικό περίβλημα του θέματος μας απασχολεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο Πρόεδρος, ε, και εμείς ε, ευχαριστούμε ε, πολύ. Νομίζω ότι προβληματιστήκαμε με το 40 ή το 14, γιατί στα αγγλικά μοιάζουν το ίδιο, λέει ο πρόεδρος. Εγώ κατάλαβα ότι είπατε 40, 40 και όχι 14, ε, γιατί το άρθρο 40 αναφέρεται στα γεωργικά. Αλλά μετά κατάλαβα ότι εννοούσατε το 114, το 114, λέει ο κύριος Χάρμπορ. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή βλέπετε ότι αρπάξαμε τον, ε, το βιβλίο με τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να το ανοίξουμε στα διάφορα άρθρα που ε, παραθέσατε για να δούμε τι ακριβώς ε, λένε. Όλες οι επιτροπές άλλωστε βασίζουν τη δουλειά τους στο βιβλίο αυτό. Σας ευχαριστώ όλους για την ε, συμβολή μας να δώσουμε την ευκαιρία στους συναδέλφους, στα μέλη της Επιτροπής να θέσουν κάποιες ερωτήσεις μετά πριν περάσουμε τον επόμενο γύρο με τους ομιλητές. Ποιος ε, έχει κάποιο ερώτημα που θέλει να θέσει στους εμπειρογνώμονες και τους ομιλητές που έχουν προσκαλέσει εδώ εν γέννη. Να ξεκινήσω εγώ αναφερόμενος στη συνεισφορά των πιστοτικών ενώσεων. Ε, είναι πολύ σημαντική η συμβολή του στη συζήτηση του όλου θέματος και θέλω να το συσχετίσω με την ύπαρξη ε, του διαφορετικού νομικού πλαισίου υπό το οποίο λειτουργούν οι πιστοτικές ενώσεις σε, κάποιες, σε όλες τις χώρες μέλη. Α, άλλωστε σε ορισμένες χώρες μέλη δεν είναι καν Ο κ. Καμπίσκη από την ε, Πολωνία μας έδωσε πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Όμως υπάρχουν και άλλα ε, θέματα με τις πιστοτικές ενώσεις που θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας. Ε, μπορούν να συμβάλλουν εδώ στο πεδίο που μας, μας απασχολεί, αλλά θα μπορούσαν να συμβάλλουν και αλλού ενδεχομένως. έτσι ώστε ο πολίτης να έχει πρόσβαση ε, σε μια πιο προσβάσιμη, να το πω έτσι, χρηματοδότηση. Και στη δική μου χώρα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ε, πρόγραμμα με συνεταιρισμούς οι οποίοι βοηθούν τους ανθρώπους να εξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις για να ξεφύγουν από τον κλειό της ανεργία. Είναι κάπως διαφορετική η οπτική γωνία που σας παρουσιάζω, είναι όμως χρήσιμο να το εξετάσουμε αυτό. Κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν και σε διαφορετικές περιπτώσεις οι πιστοτικές αυτές ενώσεις. Ο κύριος Καμίνσκι. Ε, κοιτάξτε, αυτού του είδους οι οργανισμοί παίρνουν μέρος στις δράσεις κοινωνικής συνοχής με διαφορετικούς τρόπους. Προσφέρουμε ε, προσβάσιμες υπηρεσίες ε, στις ε, διάφορες οικογένειες π.χ. που διαβιούν στην Ήπεθρο. Προσφέρονται υπηρεσίες σε διάφορους ανθρώπους που ξεκινούν τη δική τους ε, επιχείρηση, αλλά μόνο στις ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή μόνο ατομικά σε μέλη, ε, σε εταίρους που ξεκινούν μια επιχείρηση, σε ατομικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο νομικής οντότητας επιχείρησης. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό είναι η έλλειψη άμεσης πρόσβασης την υποδομή ε, ρύθμισης των πληρωμών. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα στην Πολωνία και αυτό βλέπουμε ως πρόβλημα και σε άλλες χώρες. Και τίθεται βεβαίως και το θέμα του κόστους, ειδικότερα για τις μικρές πιστοτικές ενώσεις, για τις οποίες είναι ε, δύσκολο είναι δυσβάσταχτο το κόστος ούτως ώστε να αναβαθμιστούν ως πλήρη μέλη του συστήματος ρύθμισης των πληρυθμών. Δεν υπάρχουν προβλήματα με το άνοιγμα βασικού λογαριασμού. Ο, ε, οποιουσδήποτε ε, μπορεί να γίνει μέλος μιας πιστοτικής ένωσης και να ανοίξει λογαριασμό. Προσφέρουμε επίσης δάνεια φθηνά αν θέλετε προσβάσιμα σε ανθρώπους που έχουν λευκό τραπεζικό μητρό για να το πω έτσι. Δεν είναι άλλα τα προβλήματα αυτά. Η οδηγία για την καταναλωτική πίστη στην οποία αναφερθήκατε ε, υφίσταται και στην ε, Πολωνία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό το θέμα. Δεν, ε, δεν παραβλέπουμε την οδηγία αυτή, συμμορφωνόμαστε πλήρως, εντασσόμαστε στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και θεωρούμε ότι προσφέρουμε πολλά ωφέλη στα μέλη μας. Ωστόσο κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο δημοφιλές σε ορισμένες χώρες, αλλά θα πρέπει να το τονίσω, είναι το εξής ένα τεράστιο κομμάτι της αγοράς δεν είναι καθόλου ρυθμισμένο. Όσοι δανείζουν χρήματα ε, είναι πολύ συχνά διαφορετικές επιχειρήσεις που παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες και αξιοποιούν αυτή την κατάσταση κοινωνικού αξοπλισμού για να βγάλουν χρήματα, να κερδοσκοπήσουν σε βάρος των φτωχών. Και αυτό το παρατηρούμε στην Πολωνία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδεχομένω και σε άλλε χώρε ενδεχομένω επίση. Στην Πολωνία λοιπόν αυτά τα θεσμικά όργανα δεν έχουν καμία υποπτία, δεν ρυθμίζονται από πουθενά, δεν ακολουθούν ε, τους κανόνες ή αν θέλετε μπορούν να ε, διαφύγουν, να διαλάθουν ε, τις προσοχής της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη, για παράδειγμα και είναι ένα ε, πρόβλημα που πρέπει να εντοπίσουμε. Τώρα, ως προς τις διάφορες χώρες, ενδεχομένως υπάρχει ένα πρόβλημα έλλειψης στρατηγικής ε, οικονομικής εκπαίδευσης. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται καθόλου να χαράξει στρατηγική για την εκπαίδευση ε, επί των χρηματοοικονομικών και των οικονομικών των πολιτών. Δεν θεωρούν ότι είναι... Ε, σημαντικό το θέμα αυτό οι κυβερνήσεις. Αυτά όλα είναι κάποια από τα βασικά προβλήματα. Ο Πρόεδρος, βεβαίως μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στο κείμενό μας. Ο κύριος Σμιτ και μετά η κυρία Γκέμπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσοι δεν χρειάζονται τραπεζικό λογαριασμό είναι οι άνθρωποι για τους οποίους μιλούμε. Λέει αυτό το ε, προσχέδιο κειμένου εδώ ότι 5 ή 6 ή 7% είναι ε, το ποσοστό στην Πολωνία που δεν το επιθυμεί, δεν επιθυμεί να έχει τραπεζικό λογαριασμό ή και πιο υψηλό ε, ποσοστό είναι αυτό. Άλλοι όμως λένε ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκο να έχει τραπεζικό λογαριασμό και αρνείται να τον έχει. Γι' αυτό δεν θέλει να έχει τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να επικεντρωθούμε. Και το λέω αυτό κύριε Πρόεδρε, διότι ε, προηγουμένως ε, κάνατε αυτή την παρατήρηση ότι μπορεί, μπορεί ενδεχομένως ο τομέας να αυτορυθμιστεί. Δεν το έχει πράξει όμως και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν το έχει κάνει. Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να το κάνουμε εξαιρετικά περίπλοκο. Ξέρετε, έχουμε την τάση εμείς εδώ να περιπλέκουμε πολύ τα πράγματα και κατά τη δική μου άποψη δεν μιλώ για τη χορήγηση πίστοση στον κόσμο. Ο καθηγητής κύριος Ράιφνερ μίλησε για το ποσοστό χρέους, για τους χρεωμένους πελάτες οι οποίοι χρειάζονται ε, πρόσβαση σε ρευστότητα. Αν εγώ ήμουν τραπεζίτης θα ε, αρνιόμουν και δεν θα τους έδινα, ε, δεν θα τους άνοιγα καινούριο λογαριασμό. Βασικό μου ένστικτο όμως είναι το εξής. Εάν κάθε πολίτη στην Ευρώπη θέλει ένα τραπεζικό λογαριασμό, τότε θα πρέπει να τον έχει. Όχι πίστοση, όχι πίστοση προς Θεού, αλλά τραπεζικό λογαριασμό. Εάν συζητήσουμε ε, επ' αυτής της βάσης ε, θα περιπλέξουμε πάρα πολύ τα πράγματα και δεν θα καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα. Ο Πρόεδρος, να δώσω το λόγο στην κυρία Γκέμπχαρτ και μετά στον κύριο ε, ή ο, από τους δύο θέλει. Όποιος από τους δύο θέλει ας μιλήσει πρώτος. Ο κύριος Κλούιτε. Ευχαριστώ πολύ. Δυο ερωτήσεις έχω ιδιαίτερα μετά που, από αυτά που είπε ο Λεσμίτ Και εγώ πιστεύω ότι βεβαίως πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, ε, πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό για ε, να μπορεί κανείς να κάνει ηλεκτρονικές ε, πληρωμές και αλλά όχι πίστοση. Το επόμενο ερώτημα, λοιπόν, το τεχνικό ερώτημα που τίθεται τώρα και το οποίο συνεχώς προβάλλουν οι εκπρόσωποι των τραπεζών είναι το εξής πρέπει να υπάρχει μια τραπεζική κάρτα με την οποία να μπορεί κανείς να πληρώνει χωρίς όμως να υπερχρεώνεται. Έχετε, υπάρχει απάντηση γι' αυτό, σε αυτό θα με ενδιέφερε πραγματικά να ακούσω τι γνώμη έχουν οι τράπεζες. Ε, οι τράπεζες δεν θέλουν υπερανάληψη, ναι, αλλά μπορούν να φτιάξουν μια κάρτα με την οποία να πληρώνει κανεί, αλλά να μην γίνεται υπερανάληψη, Να, μην, να υπάρχει, να σταματάει η κάρτα να λειτουργεί άμα φτάσει κανεί στο όριο του λογαριασμού. Πού βλέπετε, ε, τι γίνεται αποδεκτό τι μπορείτε να δεχτείτε, τι δεν μπορείτε να δεχτείτε. Τεχνικά είναι εφικτό αυτό που λέω εγώ. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα ένα συνάδελφος από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων μου είπε ότι ναι και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει πρόβλημα. Α, αλλά ε, μάλλον δεν θα μπορούσε ε, καν, δεν θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές οι credit unions σε εκείνη τη χώρα ή και γιατί διότι κατά κύριο λόγο δεν μπορούν δεν μπορεί να ρυθμιστεί ο κλάδος να ρυθμιστούν τα ιδρύματα αυτά τα, οι συνεταιρισμοί αυτοί Ευχαριστώ πολύ να επισύρω την προσοχή στο στο τι συζητούμε, να μην αποπροσανατολίζουμε τη συζήτηση. Ε, Τώρα εδώ μπαίνει θέμα υπερχρέωσης των συμπολιτών μας ε, και τι θα κάνουμε με το πρόβλημα της υπερχρέωσης. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο αυτό που κουβεντιάζουμε εδώ. Η πρόσβαση σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Δεν ξεχνούμε και δεν αναγνωρούμε το γεγονός ότι θα μπορούσε κανείς να υπερχρεωθεί πιο εύκολα μέσω ενό τραπεζικού οργανισμού ε, λογαριασμού τι να πω αλλά είναι άλλο θέμα αυτό από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια ερωτήματα κύριο Καμίνσκι και την κυρία Φίλη να ρωτήσω κι εγώ πως μπορούμε να φανταστούμε να κάποια εργαλεία, κατά πόσο μπορούμε να φτιάξουμε δηλαδή κάποια εργαλεία τα οποία μέσω και του βασικού αυτού τραπεζικού λογαριασμού θα εκπαιδεύσουν τους συμπολίτε μας οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν ε, τα χρήματά τους. Στην Αυστρία ε, υπάρχει μια... Ένα ταμιευτήριο, ένα είδο ταμιευτήριο, ένα τέτοιο οργανισμό που κάνει τέτοιου είδου προσπάθειε. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να ζητήσω από τους εμπειρογνώμονες να απαντήσουν. Να ξεκινήσω από την κυρία Φίλη και στη συνέχεια από τον κύριο Καμίνσκι. Αλλά ένα σύντομο ε, σχόλιο από όλους εσάς ε, για όλα αυτά που ακούσατε μέχρι αυτή τη στιγμή. Κύριε Φίλη, θέλετε μήπως να ξεκινήσετε. Ναι κύριε Πρόεδρε, ως προς τις διαδικτυακές πληρωμές και για ποια ε, κάρτα μιλούμε. Εμείς μιλούμε για τη χρεωστική κάρτα. Αυτή πρέπει να είναι μέρος του βασικού πακέτου και βεβαίως όχι η πιστοτική κάρτα. Εάν δεν υπάρχει χρήματα στο λογαριασμό, δεν μπορεί κανείς με τη χρεωστική κάρτα να κάνει καμία αγορά. Τώρα, ως προς την υπερανάληψη. Ανέφερα την υπερανάληψη ως δυνατότητα, αλλά να μην είναι αυτή μέρος του βασικού πακέτου που θα ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε να συζητηθεί ενδεχομένω σε εθνικό επίπεδο για όσε χώρε το επιθυμούν. Να προβλέψουμε δηλαδή αυστηρές προϋποθέσεις και όρια. Ε, η ιδέα είναι για την υπερανάληψη να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη. Δεν ζητούμε να ε, αποτελέσει μέρος του βασικού ευρωπαϊκού πακέτου. Και να σχολιάσω το θέμα της χρεωστικής κάρτας για τις πληρωμές στο διαδίκτυο. Ένα άλλο πρόβλημα που τίθεται είναι το εξής. Μεγάλο μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν δέχεται παρά μόνο πιστοτικές κάρτες. Άρα θα πρέπει να ζητήσουμε και από τους ε, διαδικτυακούς εμπορευόμενους να διευρύνουν τα μέσα πληρωμών που δέχονται και κυρίως μιλώ για τις εθνικές διαδικτυακές τοποθεσίες. Ε, από δικής μας πλευράς δεν ζητούμε να διευρυθούν οι δυνατότητες πρόσβασης στην πίστη, στην πίστοση μάλλον. Αυτό που λέμε είναι ότι χωρίς βασικό λογαριασμό δυσκολεύεται κανείς να έχει πρόσβαση στις λοιπές τραπεζικές υπηρεσίες, ούτε στην πίστοση ούτε στην ασφάλιση αν θέλετε, ούτε και σε διάφορες άλλες. Δεν κάνω το συσχετισμό. Χωρίς βασικό λογαριασμό όμως κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην πίστοση. Από εκεί και πέρα, όταν θα καθορίσουμε το περιεχόμενο του βασικού ευρωπαϊκού πακέτου, Ίσως δεν είναι απαραίτητο να προκαθοριστούν τα μέσα πληρωμών που αναγκαστικά θα αποτελέσουν μέρος του βασικού ε, πακέτου. Πρέπει όμως να καθοριστεί η λειτουργικότητα. Τι να μπορεί να κάνει κανείς με αυτό το πακέτο, δηλαδή να κάνει πληρωμές, να ε, ε, κάνει ανάληψη χρημάτων και ούτω καθεξής. Αυτά είναι το βασικό πακέτο που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ο Πρόεδρος. Συμφωνούμε με αυτόν τον ορισμό του βασικού λογαριασμού λέει ε, ο κύριος Καμίνσκι δεν θα δημιουργήσει αυτό ούτε στην Πολωνία, ούτε στην Ιρλανδία, ούτε στον Ηνωμένο Βασίλειο, πόσο μάλλον μετά την ε, πρόσφατη νομοθεσία που έχει υιοθετηθεί στην ε, τελευταία αυτή χώρα. Τώρα σε άλλες χώρες, στη Ρουμανία, στην Εσθονία για παράδειγμα, ίσως ο κανόνας αυτός θα ήταν ε, πρόβλημα. Είναι ανάγκη να αλλάξει η νομοθεσία στις χώρες αυτές. Αλλά δεν ξέρω πώς ε, μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα, η υπάρχει σύνδεση μεταξύ βασικού λογαριασμού και συμβουλών κατάρτισης και ε, συνοδείας αν θέλετε ε, προπόνησης εντός εισαγωγικών. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στις πιστοτικές μας ενώσεις. Δηλαδή να έχουμε ενημερωτικές εκστρατείες. Να διοργανώνουμε διάφορες δραστηριότητες σε διάφορα επίπεδα. Τα υποκαταστήματά μας βρίσκονται ε, ακόμα και σε πολύ μικρές πόλεις, σε περιοχές που δεν έχουν τράπεζες, όπου η μοναδική πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες γίνεται μόνο μέσω του υποκαταστήματος της πιστωτικής μας ένωσης. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα από τη δική μας σκοπιά. Δεν ξέρω όμως αν είναι εφικτό ε, και για τις εμπορικές τράπεζες. Θα μπορούσαμε να στήσουμε από τις εμπορικές τράπεζες να προσφέρουν δωρεάν συμβουλές στους ε, πελάτες τους και να έχουν ανεξάρτητη ε, κατάρτιση και ανεξάρτητη παροχή συμβουλών. Πολύ δύσκολα βέβαια θα κάνουν κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι είναι ε, εφικτό αυτό. Καθηγητή, καθηγητά κύριε Ράιφνερ, λέει ο πρόεδρος, θέλετε και εσείς να σχολιάσετε. Κοιτάξτε, εδώ συζητάμε τώρα για πληρωμές χωρίς πίστοση. Δεν λειτουργεί και πολύ εύκολο αυτό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δώσουμε πίστοση, αλλά από εκεί και πέρα να δώσουμε στους πιστώσες, στους πιστωτές, να, τη δυνατότητα να έχουν ε, πρόσβαση πλέον αυτή στους ε, λογαριασμούς. Γι' αυτό τα πράγματα είναι δύσκολα ε, και γι' αυτό ίσως α, ε, γι' αυτό ίσως δεν ενδιαφέρει δεν λειτουργούν και αυτοί οι βασικοί λογαριασμοί πολύ καλά και για να είμαι ειλικρινής γι' αυτό ε, δίνονται και αυτές οι τηλεφωνικές πιστώσεις όπως ξέρετε ότι δίνονται και στη Φιλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα λοιπά οι οποίοι φτωχαίνουν ακόμη περισσότερο τον κόσμο το λέω συγγνώμη που δεν θα σας αρέσει αλλά έτσι είναι Έχει τον λόγο ένα συγκεκριμένο ερώτημα στη Γερμανία υπάρχει ένα είδος προστατευμένου λογαριασμού κόντο δεν θα μπορούσε να ε, συνδυαστεί αυτό με το βασικό λογαριασμό αυτό το είδος λογαριασμού για να ε, μπορέσουμε να μην έχουμε πρόβλημα ωραία απάντηση του καθηγητή δηλαδή τι θα κάνουμε. Θα ανοίξουμε άλλον ένα λογαριασμό για αυτούς τους ανθρώπους που θα ενισχύσουμε αυτό το οποίο ονομάζω εγώ οικονομία γκέτο, οικονομία για, ειδική οικονομία, ειδικά προϊόντα για τους υπερχρωμένους. Όχι, είναι προβληματικό κάτι τέτοιο. Ε. Ακόμη και αν δεν πιστεύω ότι πρέπει να αποκλείονται από την κοινωνία μας οι φτωχότεροι. Συγγνώμη να παρεμβαίνω και εγώ γιατί είναι σοβαρό το θέμα που συζητάτε. Εκείνο το οποίο θέλουμε, δεν θέλουμε, ε, ε, δεν είναι να δημιουργήσουμε ε, εξε, ειδικούς λογαριασμούς, και ειδική οικονομία. Εκείνο που σας ενδιαφέρει είναι οι άνθρωποι να έχουν ένα λογαριασμό. Δεν μπορούν. Αυτό πρέπει να επιδιώξουμε να κάνουμε και γι' αυτό είναι και οι εμπειρογνώμονες εδώ για να μας πούν πού είναι τα προβλήματα πού ε, ε, μπλοκάρουν οι προσπάθειες αλλά επουδενή λόγο πρόκειται να δεν θέλουμε σήμερα εδώ να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να παρακάμψουμε ορισμένα πράγματα τη δημιουργία ειδικών λογαριασμών κτλ επουδενή λόγο θέλουμε κάτι τέτοιο ξέρουμε ότι υπάρχει για κάποιους πρόβλημα φρεντγκιότητας Οπότε γι' αυτό λέμε ας έχουν αυτοί οι άνθρωποι ένα βασικό λογαριασμό αλλά να είναι normal ο, ο λογαριασμός αυτός το να εφόσον η Γερμανία μου λέτε τώρα ότι φτιάχνει ειδικού λογαριασμούς για ορισμένες περιπτώσεις το κάνει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο μακάρι να επιτύχει το εγχείρημα και να μην αποτύχει Σίγουρα είναι ένα σημείο στο οποίο θα επανέλθουμε. Θέλω να ακούσω τον κύριο Ντέμπερκ και έχουμε και άλλους τρεις εκλεκτούς εμπειρογνώμους περίπου να μας μιλήσουν και θα έχουμε μια γενική συζήτηση στο τέλος. Κύριος Ντέμπερκ, μόλις τώρα βρήκα το άρθρο 14, εδώ συγγνώμη, το 14. Ζητώ συγγνώμη που δεν σε πρόφερα σωστά. Όπως ξέρετε, αυτό το να μιλάει κανείς με τα δόντια του είναι δανέζικη ειδικότητα. Έχω δύο τρία σχόλια στο κατά πόσο ένας προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να είναι να περιλαμβάνει και πρόσβαση σε, στην πίστη, την έκδοση δηλαδή πιστοτικής κάρτας. Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι έχουμε περάσει μια χρηματοοικονομική κρίση που σε μεγάλο βαθμό ε, πυροδοτήθηκε από την υπερβολικά εύκολη προσέγγιση στην πίστη. Νομίζω θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. στην διευθέτηση ή επιβολή στην ε, οικονομική πρόσβαση που ταυτόχρονα θα δίνει πρόσβαση και στην πίστη δεν θα πρέπει να υιοθετηθεί, τουλάχιστον από τις συνθήκες. Δεύτερο σημείο. Βλέπω πάρα, πολλές, πάρα πολλά τεχνικά και νομικά προβλήματα στον καθορισμό επακριβώς του τι εννοούμε με το πώς η πίστη σε ποιον και σε ποιον ανεξαρτήτως αξιοπιστίας, πιστοληπτικής ικανότητας, δηλαδή χρέωσή του κλπ. Αυτή είναι η δεύτερη παρατήρησή μου. Δηλαδή, νομικά και τεχνικά είναι αρκετά δύσκολο να διευθετήσουμε αυτό. Τρίτη παρατήρησή μου. Νομίζω ότι πραγματικά βρισκόμαστε στα όρια αυτού του ό,τι μπορούμε να αποκομίσουμε στις διατάξεις μας εσωτερικής αγοράς. Εάν θέλουμε ένας κανονισμός να βασίζεται στο άρθρο 114, 114 και το τονίζω, τονίζει ο μιλητής, το βρίσκω δύσκολο το πώς θα μπορούμε να συμπεριλάβουμε και την πρόσβαση σε πίστη, σε μια συγκεκριμένη, σε μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Νομίζω ότι η κυρία Γκέπχαρντ ακριβώς το επεσήμανε. Έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας από αυτή την έννοια. Πρέπει να εστιάσουμε μόνο στην πρόσβαση τραπεζικό λογαριασμό. Και αυτό μας οδηγεί στην επόμενη ομάδα ομιλητών. Γιατί θέλουμε να ρωτήσουμε ε, τα θέματα αυτά και από τη σκοπιά της ωφέλης στην εσωτερική αγορά. Με πολύ μεγάλη μου λοιπόν ευχαρίστηση σας παρουσιάζω για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, γιατί στο παρελθόν ήταν τακτικός επισκέπτης της Επιτροπής μας, υπό την αρμοδιότητά του ως Διευθυντής, τον Jim Murray ο οποίος ε, έχει προαχθεί σε νέο ρόλο ως ε, πρόεδρος του, της Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη χρηματοοικονομική συμπερίληψη. Και από εμάς ενδιαφέρεται ιδιαίτερα το θέμα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα από τον καλωσορίσουμε και πάλι. Μετά θα ακούσουμε τον Περνά Μπαγιό, ο οποίος ε, είναι ε, διευθύνων σύμβουλος του δικτύου εναλλακτικής χρηματοδότησης και της ε, ομάδας ε, χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τέλος θα ακούσουμε τον κύριο Ντέρκ Στάιν ο οποίος είναι διευθυντής του Ευρωπαϊκού ε, Δικτύου Τραπεζικής Λιανικής και πολιτικής, καταναλωτικής πολιτικής στο, στην Ένωση Γερμανικών Τραπεζών. Λοιπόν, εστέω στον τον πιο σύντομη για να έχουμε χρόνο και για συζήτηση. Καταρχάς ο Τζίμαρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με προσκαλέσατε και για τα ευγενικά συλλόγια. λόγια. Είναι ωραία που ξαναβρίσκομαι μεταξύ φίλων. Όντω έχω νέα αρμοδιότητα εδώ και κάποιε εβδομάδε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη χρηματοοικονομική ε, συμπερίληψη που ιδρύθηκε το 2010 προκειμένου να παράσχει ακριβώς προσπέλαση ε, σε τροπεζικό λογαριασμό στους πάντες, περιλαμβάνοντας βέβαια, όπως καταλάβατε, και τις διαφορετικές εναλλακτικέ. Μου προσφέρθηκε αυτή η δουλειά και χάρηκα γιατί δεν την αναλάβω. Τρει παρατηρήσει έχω να κάνω. Καταρχά, οικονομική μεγέθυνση στην ενιαία αγορά, γιατί αυτό είναι και ο βασικό στόχο αυτού του κομματιού τη συνεδρίαση. Δεύτερη παρατήρηση πάνω στους βασικούς ε, λογαριασμούς πληρωμών και σε τι θα πρέπει να αποτελείται. Και τρίτον, κατά πόσον είμαστε υπέρ μιας ε, υποχρεωτικής προσέγγισης. Συμμερίζομαι την κριτική της κυρίας και άλλων σε ό,τι αφορά την χαλαρή προσέγγιση, αλλά σίγουρα το θέμα της υποχρεωτικής προσέγγισης θα πρέπει να εκφραστεί επίσης και ελπίζω να συμφέρω σε αυτό η οικονομική υπόθεση και το κοινωνικό επιχείρημα, αν θέλετε, για τα 30 εκατομμύρια ανθρώπους και περισσότερους που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό είναι σημαντικό. Αλλά υπάρχουν και υπερασπιστικά επιχειρήματα και από πλευρά ενοποίηση τη κοινή αγορά, αλλά και οικονομική μεγέθυνση. Η οικονομική μεγέθυνση είναι καλύτερη όταν είναι, όταν είναι συμπεριληπτική, όταν οι πάντε μπορούν να συμμετάσχουν με βάση βέβαια ο καθένα των δυνατοτήτων του και η πρόσβαση στι χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε ήταν κεφαλαιόδου σημασία γι' αυτό. Επίση, χωρί να επισέρχομαι στι διάφορε περιπλοκέ των άρθρων τη συνθήκη, είναι επίση πολύ σημαντικό να υπάρχει καθολική προσέγγιση στι υπηρεσίε γενικού ενδιαφέροντο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεισφέρει σημαντικά στην μεγέθυνση του τρόπου που αναπτυσσόμεθα στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε όμω να επιτύχουμε την πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίε γενικού συμφέροντος χωρί πρόσβαση στους κατάλληλων μεθόδων πληρωμής. Η καθολική προσέγγιση θα ήταν ατελής αν δεν μπορούμε να, πληρώσουμε για τι υπηρεσίε αυτέ και δεν έχουμε τα μέσα για να το κάνουμε. Επίση, το ίδιο, μιλήσαμε για 30 εκατομμύρια, Ενδεχομένω, είναι και περισσότεροι οι πολίτες και βέβαια αυτό εξαρτάται από τη μεθοδολογία που ακολουθείται στη δημοσκόπηση και τη μέτρηση. Αλλά εν πάση αν σκεφτώ τα 30 εκατομμύρια αυτά δεν είναι όλοι ε, αβοήθητα θύματα. Πολλοί εξ αυτών, ίσως και οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει πάρα πολλοί, αποτελούν το δυναμικό για καινοτομία, για επιχειρήν, για συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά εμποδίζονται από το να το κάνουν αν δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό και πλήρωση με τραπεζικού λογαριασμού. Η οικονομική μεγέθυνση δεν προέρχεται μόνο από τους κεφαλαιοκράτες ή με, με πολύ ή με αυθονία μέσω παραγωγής διάθεσή τους. Επίσης, συναρτήσεις του χρόνου έχουν αυξηθεί εκείνοι οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην τράπεζα, αλλά η με αυθονια μεσω παραγωγης διαθεση τους επισης αρτηση του χρονου εχουν αυξηθει εκεινοι οι οποιοι εχουν προσβαση στην τραπεζα αλλα η προοδος θα καταγραφεί πάρα πολύ αργά αν περιμένουμε μέχρι ότου οι τράπεζες είναι έτοιμες να παράσχουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε μεγαλύτερο αριθμό. Η μεγέθυνση θα προέλθει πολύ νωρίτερα εάν οι νωρίτερα έχουν οι περισσότεροι τραπεζικού λογαριασμού. Και στα πλαίσια τη αγορά, επίση είναι προφανέ, οι πληρωμές ε, και οι αναλήψει ε, είναι πολύπλοκες διασυνοριακά, είναι δαπανηρέ, και σε πολλέ περιπτώσει είναι και ε, ανέφικτες χωρίς πρόσβαση σε κάποιο βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Σίγουρα καλωσορίζουμε λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν θεωρούμε ότι είναι αρκετά τολμηρή. Για την πλειοψηφία των ατόμων που υποφέρουν ιδιαίτερα από τον οικονομικό αποκλεισμό, η ικανότητα να καταθέτουν και να κάνουν αναλήψεις μετρητών παραμένει πολύ σημαντικό στοιχείο για πάρα πολύ καιρό. Θα πρέπει να το εξετάσουμε λοιπόν αυτό, σε πώς έχουν πρόσβαση σε αυτόματα μηχανήματα ή διαθετήσεις που υπάρχουν για καταθέσεις. Και η οδηγία είναι ατελή στο σημείο αυτό. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία ανέφεραν άλλοι ομιλητέ για την επέκταση του βασικού τραπεζικού λογαριασμού που δεν θα αναφέρω εδώ. Κάποιοι νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο η διεθνή και η online τραπεζική συναλλαγή είναι η απάντηση. Αλλά αυτό δεν λύνει το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού στο ορατό μέλλον. Κάθε άλλο. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ όμως ανάμεσα στους χρηματοοικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένους το online banking μάλλον θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο την ψαλίδη μεταξύ αυτών που έχουν τραπεζικό λογαριασμό, των εχόντων, κατεχόντων και των μη εχόντων και κατεχόντων. Βέβαια όλο αυτό δεν είναι σφάλμα των τραπεζών κατά κάποιο τρόπο. Πρέπει να είναι διαθέσιμο όχι μόνο τραπεζικό λογαριασμό πληρωμή, αλλά πρέπει να ληφθούν ε, βήματα για αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό λογαριασμό. Πρέπει να γίνουν βήματα λοιπόν για να φτάσουμε τους ε, πλέον αποκλεισμένου, είτε μέσω των δημόσιων αρχών, των μη κυβερνητικών οργανισμών, αλλά και από τράπεζε. Δεν πρέπει να κάθονται παθητικά και να περιμένουν, αλλά επίση θα πρέπει να προσπαθούν να ενθαρρύνουν του αποκλεισμένου. Και επίση οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα πρέπει να είναι πιο ορατοί, πιο προσιτοί, ακριβώ για να υπάρξει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Τέλος, το θέμα του κατά πόσο πρέπει να είναι υποχρεωτική για προσέγγιση. Όχι με το, για το, με το σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά για μια πιο δεσμευτική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη και θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερε συνθήκες τους. Στην, ε, ε, στην έκθεση επιπτώσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλούν για έναν κανονισμό πλαίσιο. Δεν πρόκειται να επισέλθω να σου πω σε ποιο άρθρο αναφέρεται, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι απαραίτητο, κάτι τέτοιο αναφέρεται. Καταρχά, οι τράπεζε δεν πρόκειται να, κερδο, να έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία από του βασικού τροπικού λογαριασμού για κάποιο διάστημα. σω να είναι πολύ πιο κερδοφόρε από ό,τι το ομολογούν αυτή τη στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν παρέχουν λογαριασμού σε πολύ μικρό περιθώριο κέρδου, δεν είναι η πλέον κερδοφόρο δραστηριότητά του. Έτσι λοιπόν ένα μη δεσμευτικό εργαλείο κατά, κατά κάποια πιθανότητα θα είναι αναποτελεσματικό και διακινδυνεύει ε, ίσως να προάγει, ε, να υποθάλψει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Οι διάφορες εστάσεις και το ήπιο δίκαιο δεν λειτουργούν σε αυτή την περίπτωση. Για παράδειγμα, σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρωμής, με πληροφόρησης για στεγαστικά, σε σχέση με τις ε, προμήθειες των τραπεζών και πιο λίπιο πρόσφατο σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις. Αντίστοιχα, εάν ακολουθήσουμε την ήπια προσέγγιση θα είναι αναποτελεσματικό το μέτρο. Εξεπλάγει από διάφορου ε, συναδέλφους που άκουσα και γίνεται μαρτυρία από την έκθεση επιπτώσεων, όπου οι Γερμανοί πολίτες λένε ότι υπήρξε το 1996 προσέγγιση ήπιου δικαίου πριν από 16 χρόνια, αλλά δεν πέτυχε τους στόχους της. Επίσης επισήμαναν κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι υπάρχει κάποιο ομόσπονδο κρατήδιο που για κάποιους πολύπλοκους λόγους ε, όντως έχει ακολουθήσει δεσμευτική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού. Σε εκείνα τα ομόσπονδα κρατήρια που υπήρχε αυτό υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με τα ε, ομόσπονδα κρατήρια όπου δεν υπάρχει τέτοιου είδους διευθέτηση, έχει ακολουθηθεί το ήπιο δίκαιο. Οι συστάσεις λοιπόν και το μαλακό απαλό δίκαιο έχουν, λειτουργούν ορισμένε φορές με περιορισμένα αποτελέσματα σε κάποια κράτη-μέλη συγκεκριμένου τομεί. Έχει λειτουργήσει καλά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά δεν μπορούν αυτά τα αποτελέσματα να επαναληφθούν σε όλα τα κράτη-μέλη γιατί υπάρχουν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις και παραδόσεις απέναντι στο ήπιο δίκαιο της συστάσης και τους κώδικες εντολογίας των διαφορετικών κρατών μελών. Δεσμευτικά λοιπόν μέτρα μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί όλα τα κράτη υπόκεινται στο κράτος δικαίου. Δεσμευτικά μέτρα επίσης πρημοδοτούνται από αυτούς που είναι πολύ πιο πεπισμένοι, πολύ πιο συνδυσμένοι να εργάζονται με τους κοινωνικά οικονομικά αποκλεισμένους. Ας πούμε για παράδειγμα ότι είμαι ακόμα μεγαλύτερος, γυρεότερος και από ότι είμαι, ότι έχω τραπεζικό λογαριασμό, πάω σε μια τράπεζα, ο διευθυντής βλέπει σαφέστατα ότι δεν πρόκειται να του προσφέρω και πολύ μεγάλο κέρδος, δεν θα είμαι πηγή μεγάλου εισοδήματος για την τράπεζα, δεν είμαι εκεί ιδιαίτερα ελκυστικός. Πώς μπορώ να πείσω λοιπόν το διευθυντή της τράπεζας ότι θα πρέπει να μου ανοίξει κάποιο λογαριασμό. Δεν μπορώ να πω, ο, απαιτείται Πρέπει να το κάνετε γιατί υπάρχει σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Φρυξέλλες. Δεν νομίζω θα ήταν και πολύ ε, αποτελεσματική η προσέγγιση. Ή θα μπορούσα να πω υπάρχει νόμος. Αυτό θα ήταν αποτελεσματικό. Επανερχόμενος όμως στο θέμα των μαρτυριών, υπήρξαν τόσες πολλές συστάσεις στο πεδίο αυτό που έχουν ακολουθηθεί με αποδεσμευτικά μέτρα. Η μαρτυρία λοιπόν είναι πασιφανής. Δεν καταλαβαίνω την ε, δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ακολουθεί το θέμα της σύστασης. Μοιάζει λίγο με την εμπειρία κάποιων δεύτερων γάμων που είναι ο θρίαμβος της ελπίδας ναι. σε σχέση με την εμπειρία. Εν συνόψη λοιπόν, ο βασικός τραπεζικός λογαριασμός θα συνεισφέρει στην μεγέθυνση, τη συμπερίληψη, στην πραγματική ενιαία αγορά και τη λειτουργία του εμπορίου συνοριακά. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένε διατάξεις για να ενισχύσουμε το βασικό σύστημα πληρωμής λογαριασμού, να μπορέσει να προχωρήσει πολύ περισσότερο. Και τέλος, είναι το επιχείρημα, το επιχείρημα υπέρ μιας υποχρεωτικής προσέγγισης είναι σαρωτικό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινήσαμε, ξεχάσαμε να σας βάλω με το ρόλο να ξεκινήσατε και ούτως ή άλλως τα είπατε τόσο γρήγορα που σίγουρα ε, ήσταν απόλυτα ε, συνεπείς. Κύριε, Πρόεδρε, θα μιλήσω εκ μέρους των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος είναι ε, στην, ε, σε ό,τι αφορά την, ε, την Ένωση την οποία εκπροσωπώ να παρέχουμε γνωμοδοτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παρέχουμε συμβουλές και πολιτικές, να δούμε όταν υπάρχουν βασικά επιχειρήματα Προστικοποιούμε πληροφορίε για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με στα αντιπροσωπευτικά όργανα σε επίπεδο ευρωπαϊκό και, και εθνικό. Η FSUG έχει 10, 20 μέλη που εκπροσωπούν ε, τα συμφέροντα καταναλωτών, μικροεπενδυτών και επιχειρήσεων. Και είμαστε εμπειρογνώμονες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εκ μέρους της ομάδας ε, χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πέρσι τον Ιούλιο η FSUG απέστειλε στον πρόεδρο της Επιτροπής Μπαρόζο και στον Επίτροπο Μπαρνιέ εκφράζοντας σημαντικές ανησυχίες σε σχέση με την ε, πρόταση, πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση οδηγίας για τις μετακοινωνικές υπηρεσίες. Οι αποφάσεις φέγονται αντιφαντικές όταν είχαν, αφού πλέον είχαν εντοπιστεί σαν βασικό σημείο για την ε, αύξηση της μεγέθυνσης και πρέπει να και είχαν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν του 2011. Δύο επιχειρήματα παρουσιάστηκαν. Πολλέ μελέτε καταλήγουν ότι το να έχει κανεί πρόσβαση σε βασικέ χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε είναι ζωτική σημασία για να ενταχθούν οι πολίτε στην κοινωνία και να πάψουν να περιθωριοποιημένοι. Είναι το πρώτο βήμα για μια καλή χρηματοοικονομική συμπερίληψη που ορίζεται από την έκθεση Ευρωπαϊκή Ένωση του 2008 ως το δικαίωμα κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση στην και χρήση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων στην βασική αγορά, στην αγορά κυρίου κορμού και όχι κορμού υπηρεσίων δηλαδή και προϊόντων που θα έχουν δημιουργηθεί για τις ανάγκες τους και θα τους δίνουν τη δυνατότητα να διάγουν μια φυσιολογική κοινωνική ζωή στην κοινωνία στην οποία ανήκουν η χρηματοοικονομικός αποκλεισμός συνδέεται πολύ στενά και άμεσα με τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Επιπροσθέτως, είναι βασικά θέματα του, της ε, συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Τα βασικά δικαιώματα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια διακυβεύονται εδώ, υπό την έννοια του, όπως τις θέσεις που θέλει η Γενική Διεύθυνση. Είναι θέματα αξιοπρέπειας, προσωπικής ε, ζωής, και η κατήσχηση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένων βέβαια μειονοτήτων. Το δεύτερο σημείο είναι η αμαγέθυνση της εσωτερικής αγοράς. Ο χρηματοοικονομικός ε, αποκλεισμός μπορεί να συνιστά εμπόδιο στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται στο πρόγραμμα δράσης το οποίο είχε θετηθεί το 1999 ότι ε, η χρηματοοικονομική συμπερίληψη είναι θεμελιώδης για να έχουμε μια ενοποιημένη εσωτερική αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επίσης, στο στην Λευκή Χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2000-2010 τονίζεται ότι η πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό είναι το βασικό εφαλτήριο για τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές και για τους πολίτες να συμμετέχουν στην αγορά και την κοινωνία. Και τέλος, στην ανακοίνωση του περασμένου Απριλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την πράξη ενιαίας αγοράς όπου αναφέρεται στην ανικένωση, ότι θα πρέπει μέχρι το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μέτρα που θα εξασφαλίζουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πλαίσιο που θα επιτρέπει στους πάντες να επιτελούν το καθήκον τους. Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν είναι όλοι οι πολίτε ε, ικανοί να συμμετέχουν ενεργά στην ενιαία αγορά, να έχουν πρόσβαση δηλαδή σε βασικέ χρηματονομικές υπηρεσίε που έγινε βασική προπόθεση για την συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Κάτι τέτοιο δεν είναι προσιτό σε όλου. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια πρωτοβουλία που θα αφορά την πρόσβαση σε έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών σε λογικό κόστο για όλου του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. κατά την άποψη της FSUG, της ομάδας που εκπροσωπώ, μια απλή σύσταση δεν είναι σωστή λύση. Πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικό μέτρο όσο θα ήταν μια νομοθετική πρόταση για να επιληθεί το πρόβλημα αυτό στους, και να επιλύσει το πρόβλημα 30 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρώπης. το μαλακό δίκαιο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις παραβίασης βασικών δικαιωμάτων των πολιτών. Ήδη το 2001 η, η Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτικών ε, Ενώσεων αναποφάνθηκαν ότι το ήπιο δίκαιο δεν μπορεί να επιλύσει βασικές καταστάσεις. οι, αυτοκανανιστικά μέτρα προκαλούν ανισότητα των κρατομελών. Ως εκ τούτου οι πολίτε σε κάποια κράτη-μέλη είναι χρηματοοικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένοι. Το, το μαλακό δίκαιο δεν είναι το κατάλληλο για την καταπολέμηση της κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη. Όπω αναφέρθηκε και προηγουμένω, το να μην έχουμε πρόσβαση σε έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να κάνει να καταταστήσει ανέφικτες και απροσπέλαστες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Είναι υπερβολικά χρονοβόρες και ε, πανηρές ε, και ίσως κάποια δουλειά να γίνεται πολύ δύσκολη με δεδομένο ότι περισσότεροι μισθοί πληρώνονται, καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πλέον να έχει συνειδητοποιήσει το 2012 ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολιτές, αναθεωρώντας τη θέση της. Για καθιστώντας εφικτή την, πρόση, την προσπέλαση ε, όλων σε τραπεζικό λογαριασμό. Ευχαριστώ τον κύριο Μπαγιό, λέει ο πρόεδρος. Τελευταίος ομιλητής θα είναι ο κύριος Στάιν. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, πρόεδρο Μάλκορμ για την πρόσκληση εδώ. Θα κάνω μια σύντομη ε, παρουσίαση για να υπάρχει λίγο χρόνος να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα στην ε, Γερμανία το μεγάλο εγχείρημα εδώ είναι η αυτορύθμιση των ε, διαφόρων κλάδων. Στην ε, Γερμανία από το 1995 συνειδητοποιήσαμε την, το, τα προτερήματα του να έχει ένα βασικό τραπεζικό ο, λογαριασμό ο, ο κάθε ένας. Αυτό το χειροκόντο γύρω κόντο Φιωγίδερμαν, ήταν ένα σύνθημα το οποίο πραγματικά ε, το οποίο πραγματικά ε, ξεσήκωσε τον κόσμο και οδήγησε αυτή τη στιγμή σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια τέτοιους καταθετικούς ε, λογαριασμούς που ίσως να μην υπήρχαν πριν. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ένας διαμοσολαβητής, ένας ombudsman για τα θέματα τα οποία μπορεί να προκύπτουν σχετικά. Αυτό μέσα στα πλαίσια μιας αυτορύθμισης του κλάδου. Η υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα ή το ρίσκο αν θέλετε της κατάχρησης και ακόμη και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μπορεί κάποιος να ζητήσει να έχει ένα τέτοιο λογαριασμό ή από εκεί και πέρα μπορεί ο κάτοχος του λογαριασμού να μην έχει πλέον ε, έσοδα ή να μην μπορεί να διαχειριστεί τα έσοδά του κτλ. Εάν και οποιαδήποτε τράπεζα θέλει να απορρίψει το αίτημα ενός ε, πελάτου για τέτοιου είδους απλό βασικό λογαριασμό τότε πρέπει να το κάνει γραπτά και οι 5% των παραπώνων σε σχέση με τα σε, σε σχέση με τα, τις υποθέσεις που πάνε στον Ombudsman, σε αυτόν τον διαμεσολαβητή, 266 ε, από τις 5.300 υποθέσεις σχετίζονταν με αυτόν τον βασικό λογαριασμό για τον καθένα, όπως τον λέμε. Βεβαίω, όπω σα είπα υπάρχουν, υπάρχουν και οι περιπτώσει όπου κάποιο δεν μπορεί να διαχειριστεί τα χρήματά του και δημιουργούνται προβλήματα αλλά θεωρούμε ότι είναι καλύτερα να υπάρχει ένα λογαριασμό για κάθε ένα παρά να βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρίσκονται άλλε χώρε με πολύ ψηλά ποσοστά πολιτών χωρίς λογαριασμό καθόλου. το γεγονός ότι σε πάρα πολλές χώρες ε, νομοθετικά επιβάλλεται η δυνατότητα πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό ε, δείχνει ότι οι χώρες αυτές έχουν πιστεί για την ανάγκη ενός τέτοιου βασικού ε, λογαριασμού. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα νομοθέτημα ή ένας κανονισμός αν θέλετε, μια ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί πραγματικά είμαστε πεπισμένοι ότι χρειάζεται να έχει ο κάθε πολίτης ένα λογαριασμό. Βεβαίως θα, και βεβαίως θα πρέπει να οριστούν ε, κάποια ελάχιστε υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από το λογαριασμό αυτό κατάθεση, ανάληψη μετρητά από τα, ATMs ε, κλπ δεν είναι τελικά ανησυμεταχείριση του Ευρωπαίου πολίτη να μπορεί να έχει όχι λογαριασμό ανάλογα με τη χώρα στην οποία κατοικεί ή στην οποία μεταβαίνει. Ε, θα πρέπει δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται να ε, επιβληθούν συγκεκριμένοι κανόνες για, το, για τα τέλη, τα τραπεζικά που θα υπάρχουν για μας. Στην ε, Γερμανία ο, ο λογαριασμός αυτός ο βασικός είναι ο ίδιος λογαριασμός όπως έχουν όλοι οι πολίτες και χρεώνονται τα τέλη κανονικά. Αλλά εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει νομοθετική ε, πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι ήταν σαφέστατη η παρουσίασή σας και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν. Ε, προγραμματίζουμε να κλείσουμε την ακρόαση στις 6.30 ακριβώς. Θα δώσω τώρα το λόγο για να δεχθείτε ερωτήσεις από τα μέλη, αλλά βεβαίως και οι υπόλοιποι ομιλητές μπορούν να παρέμβουν. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάρεϊ για να απαντήσει στην πρόταση του κυρίου Στάιν κατά πόσο το σύστημα της αυτορύθμισης ε, θα μπορούσε να είναι λειτουργικό. Ε, ποιος θα ήθελε λοιπόν να το σχολιάσει. Ο κύριος Μάρεϊ πρώτα και μετά βεβαίως και οι συγητές. Ο κύριος Σμιτ, η κυρία Βαγνιό. Ο κύριος Μάγερ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τρία θέματα παρόλο που υπάρχουν πολλά μα πολλά ερωτηματικά εδώ. Αυτοί οι λογαριασμοί για ποιον φτιάχνονται, για ποιον ανοίγουν, για τους... Θα υπάρχουν πρώτον οι φτωχοί αν θέλετε της συγκεκριμένης χώρας, αλλά όλο και περισσότεροι θα είναι ξένοι Ευρωπαίοι πολίτες κατά πάσα πιθανότητα που θα έρχονται για σπουδές ή που θα έρχονται για δουλειά. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι το εξής. Τι πόσους λογαριασμούς μπορεί να έχει ο κάθε πολίτης στη χώρα μου μπορώ να έχω ένα στη χώρα που σπουδάζω άλλον έναν στη χώρα που πάω να δουλέψω άλλον έναν Τέλος πάντων, δεύτερο ερώτημα. Επισφάλειες υπάρχουν σε όλους τους λογαριασμούς. Δεν είναι η ρίσκα αναλαμβάνει η τράπεζα έτσι κι αλλιώς το ε, ακόμη είτε μπορώ είτε δεν μπορώ να κάνω ε, υπερανάληψη και υπάρχουν ε, αν, θέλετε πάντα προϊόντα στο ίντερνετ το οποίο, τα οποία όπως ελέγχθησαν ελέγχθη κοστίζουν φτηνότερα, σου έχουν, ε, χάνουν έκπτωση. ε, επειδή πουλούνται στο ίντερνετ μπορώ να αγοράσω τα προϊόντα αυτά τι απόφαση παίρνω εγώ σαν πολίτη θέλω να, ε, να έχω ένα λογαριασμό για να χρησι, τον χρησιμοποιώ για το διαδίκτυο ε, τρίτο ερώτημα ε, από την πείρα, από την εμπειρία μάλλον που είχαμε μέχρι τώρα. Ε, ακούσαμε να υπάρχουν συστάσεις ε, να υπάρχουν συστάσεις ε, οι οποίες όμως δεν κάνουν τίποτα σαν αποτέλεσμα ε, μήπως πρέπει να εφαρμοστεί περισσότερη πίεση στα κράτη-μέλη ή θα πρέπει να χτυπήσουμε τα κράτη-μέλη για αυτό ρύθμιση. Το παράδειγμα της Γερμανίας, παραδείγματος χάριν. Ε, Βεβαίως πάντα θα υπάρχει η, το ρίσκο της απάτης. Ε, θα μπορούσαν όμως να βρεθούν τρόποι να μην, να αποφεύγονται οι απάτες. Λοιπόν, ε, αυτά είναι τα ερωτήματά μου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μανιού. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχουμε ακούσει πολλά πράγματα και θα ήθελα γι' αυτό να ευχαριστήσω. Oui, après tout ce que nous... Ακούσαμε λοιπόν πολλά πράγματα και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ειδικού πυρογνώμονες που α, μας εξήγησαν αυτά μας εξήγησαν. λίγο στο εξή συμπέρασμα. Ε, επειδή με τρόμαξαν τα νούμερα για τον οικονομικό αποκλεισμό και όχι μόνο γιατί είναι και κοινωνικός αποκλεισμός ε. αν δεν έχει κανείς τραπεζικό λογαριασμό κάπου αποκλείεται και όχι μόνο από την οικονομία αλλά και από την κοινωνία πράγματι λοιπόν τρόμαξα με την ε, ε, με τα νούμερα αυτά και ευχαριστώ και τον εμπειρογνώμονο μα εξήγησε το άρθρο 14 και το άρθρο 16 γιατί και εγώ είχα την εντύπωση ότι όλοι μπορούν να έχουν έναν α, λογαριασμό άμα θέλουν πολύ βασικό Τώρα από εκεί και πέρα τι να κάνουμε, να πιέσουν τα κράτη-μέλη, να πιέσουμε τις τράπεζες, να το κάνουμε εδώ και χρόνια και δεν καταλήγουμε πουθενά να... Ε, ε κάποιος είπε ότι σε τελευταία ανάλυση πρόκειται περί της ανθρώπινας αξιοπρέπειας, το είπε η κυρία από το Γραφείο Καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό σε γενικέ γραμμέ φαντάζομαι ότι πρόκειται για άτομα τα οποία όντω έχουν οικονομικέ δυσκολίε. Ε, πρόκειται για τους φτωχού, οι οποίοι ε, τελικά αποκτούν και υπαρξιακό πρόβλημα θα έλεγα εγώ πέρα από οποιοδήποτε αίσθημα αποκλεισμού που μπορεί να έχουν διότι δεν υφίστανται είναι κάτι σαν τους άστεγους, οι άστεγοι που είναι στο δρόμο και, ε, ε, ε, ε ή αυτοί που δεν έχουν λογαριασμό που δεν υφίστανται στη, στην κοινωνία μας είναι αυτοί που πρέπει να μας απασχολήσουν αλλά τους άστεγους ας πούμε και του, τους βοηθούν μη κυβερνητικοί οργανισμοί οι οργανισμοί άλλοι που δεν έχουν και πολλά, πολύ μεγάλα κονδύλια. Ε, λοιπόν, μου λέτε τώρα ότι αυτοί μπορούν να βοηθήσουν και οι τράπεζες που έχουν ένα τόνο λεφτά ή ενισχύονται κάθε λίγο και λιγάκι από τους φορολογούμενους από τα κράτη-μέλη, δεν μπορούν να βοηθήσουν. Έφτασε νομίζω η στιγμή να αναλάβουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο να νομοθετήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Μάθαμε ξε, και ακούσαμε ξανά ότι η Γερμανία είναι πολύ αποτελεσματική χώρα. Σωστό αυτό. Αλλά οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι όλες το ίδιο αποτελεσματικές όπως και η Γερμανία. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζικών Ιδρυμάτων, εσείς είστε στο γερμανικό κομμάτι, κύριε Στάιν. Μπορείτε να πείστε τους συναδέλφους σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πανευρωπαϊκό επίπεδο ότι χρειάζεται να αντιγράψουμε το μοντέλο σας. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλες οι τράπεζες είναι κακές. Απλώς μας χρειάζεται να υγιής τραπεζικός κλάδος στην Ευρώπη. Λοιπόν, τι να σας πω. Προσπαθήστε να πείστε εσείς για αυτορύθμιση αλλά φαντάζομαι ότι και ο κύριος Χάρμπρο ο πρόεδρος θα μπορούσε να συμφωνήσει ότι αν δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό της αυτορύθμισης της εθελούσιας το εθελούσιου περιορισμού αν θέλετε του κλάδου ή της εθελούσιας πρωτοβουλίας της πρωτοβουλίας πρέπει να πάρθει στον κλάδο να πρέπει να αρχίσουμε να απειλούμε με νομοθεσία αλλά σε πρώτη φάση ρωτώ τον κύριο Στάιν μπορείτε να κάνετε τους συναδέλφους σας να συμπλέψουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την αυτορύθμιση. Πρόεδρος. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε το λόγο και στους τρεις εμπειρογνώμονες να απαντήσουν και θα ήθελα αν είδε ναι, δυνατόν να δώσουμε και το λόγο στο Λέ διότι ο Τζόναθεν Φουλ που ήταν εδώ ε, έφυγε γιατί δεν μπορούσε να μείνει ε, ο Λέ όμως ήταν εδώ όλο το, για όλο αυτό το διάστημα και είναι, ε, εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ασχοληθεί ε, με τα θέματα αυτά οπότε θα θέλαμε να του δώσουμε τη δυνατότητα να κάνει και αυτός κάποια σχόλια επίσης και ο κύριος Μίλλερ θα πρέπει να κάνει κάποια σχόλια θα δώσω λοιπόν λίγα λεπτά στον καθένα και μετά στην εισηγήτρια για να κλείσουμε την ακρόαση Thank you, ε, Ευχαριστώ πρόεδρε εγώ δεν είμαι πυρογνώμονας ιδιαίτερα για την γερμανική κατάσταση. Το παράρτημα, στο παράρτημα 6 όμως της μελέτης ε, αντικτύπου της Κομισιόν περιγράφει την κατάσταση στη Γερμανία ε, και από το 1995 και δόθε το ZK της, ε, τραπεζική, της Ένωσης, Τραπεζικής Ένωσης Γερμανίας ε, ασχολείται με τα θέματα αυτά, κάνει συστάσεις και το Δεκέμβρη του 2008 ε, βλέπουμε ότι ο αριθμός των αυτών που δεν έχουν ε, λογαριασμό παραμένει σε εκατοντάδες χιλιάδες. Η, η γερμανική κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι θα πρέπει ε, να συνεχίσουμε με δεσμευτικό κώδικα συμπεριφοράς ε, δεοντολογίας ο οποίος θα πρέπει να επιβάλλεται. Εγώ φοβάμαι να διαφωνήσω με τη γερμανική κυβέρνηση κύριε Πρόεδρε άμα λέει αυτά. Μάλιστα λέει ο Πρόεδρος δίκιο έχετε. κύριος Μαγιό, Μαγιό. Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να μελετήσουμε την κατάσταση στην κάθε χώρα χώρια. Άχα πολλά πράγματα να πω στη Γερμανία, αλλά η κατάσταση είναι σαφής. Σήμερα ζούμε ένα καθεστώς αυτορύθμισης εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιο είναι το αποτέλεσμα 30 εκατομμύρια άνθρωποι δίχως λογαριασμό Δεν αρκεί λοιπόν η αυτορύθμιση για να μην υπάρχουν οικονομικά αποκλεισμένοι πολίτες στην Ευρώπη. Εγώ θεωρώ ότι δεν λειτουργεί η αυτορύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα έλεγα και όλα ότι το αντίθετο ισχύει. Οι τράπεζες εδώ στο Βέλγιο από το 2003 ε, υπάρχουν, προ, γίνονται προσπάθειες για να ε, προχωρήσουν σε διάφορες κοινοτομίες και καινοτόμα προϊόντα οι τράπεζες. Κάποιες τράπεζες προσφέρουν προϊόντα εναλλακτικά προς τους καλασικούς λογαριασμούς. Ίσως λοιπόν αυτό θα πρέπει να γίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καινοτομία. Τώρα, η νομολογία εδώ και 10 χρόνια λέει ότι η πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές ε, υπηρεσίες είναι καθολική υπηρεσία. Παραδείγματο χάρη είναι η Postbank στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι τράπεζα. Ε, έχει, ε, χρησιμοποίησε αν θέλετε την ομολογία του Καστηρίου ε, και το επιχείρημα της καθολικής υπηρεσίας για να ε, πια κάνει αυτούς τους βασικούς λογαριασμούς. Από εκεί και πέρα Εκείνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε και να πούμε είναι ότι είναι δικαίωμα, δικαίωμα του Ευρω... που είναι γεγονός, δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη το να έχει έναν τραπεζικό λογαριασμό. αυτή τη στιγμή αποκλείονται αν με ενδιαφερόμαστε να τους βοηθήσουμε μπορούν να βοηθηθούν νομίζω. very much. Uh, Ja, vielleicht, ähm, Stein, πρώτα-πρώτα να απαντήσει τον κύριο Σμιτ. Κοιτάξτε εγώ, εμείς δεν θέλουμε να επιβάλλουμε το γερμανικό μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να εξάγουμε τα, αυτά που κάνουν οι γερμανικές τράπεζες ή να παραστήσουμε τους σούπερ αποτελεσματικούς. Ε, αλλά λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκείνο που μπορεί, ότι οι πολίτες έχουν κάποιο δικαίωμα ε, ε, με ε, κάποιες βασικές ε, για κάποιες βασικές ε, τραπεζικές υπηρεσίες και θα πρέπει να επιμείνει σε αυτό εγώ λέω ότι δεν χρειάζεται να νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό λέω τώρα για τον κύριο Μάρε να πω ότι υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι θα πρέπει να ε, νομοθετη, υπάρξει και ένα νομοθέτημα στη Γερμανία αλλά η κυβέρνηση της ε, ε χώρας μου λέει ότι δεν βλέπει αρι... να υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων χωρίς λογαριασμό ε, πάνω από 99% έχουν λογαριασμό στην Γερμανία σχεδόν όλοι έχουν λογαριασμούς και ένα τέτοιο νομοθέτημα δεν θα βοηθάει αυτό το πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό ίσως όμως θα βοηθάγε στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Σουηδία ή στις Χώρε χώρες που όπου οι άνθρωποι δεν έχουν, υπάρχει μεγάλο ποσοστό πολιτών που δεν έχουν λογαριασμούς. Κύριε Μιλουέλ, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, ένα μικρό θέμα θα ήθελα να θέσω. Μιλάμε για οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Όμως, το πρόβλημα που δημιουργείται λόγω κινητικότητας είναι διαφορετικό. Ε, ίστους λείπουν ε, από αυτούς που ταξιδεύουν και πάνε σε άλλη χώρα το προ... για αυτούς το πρόβλημα είναι κυρίως πρόβλημα χαρτιών αποδεικτικών για το που ζουν που μένουν, τι κάνουν και τα λοιπά στη Σουηδία ζητείται να υπάρχει, να είναι κανείς κάτοικος για κάποιο χρονικό διάστημα. Πόσο, δύο μέρες, δύο εβδομάδες, δύο μήνες, δύο χρόνια. Λοιπόν, αυτό εκεί οι, οι ήδη επιβληθέντες κανόνες και νόμοι δεν μπορούν να εφαρμοστούν σωστά και ίσως εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Πρόεδρος, όντως ίσως η διαφορετική εφαρμογή ή η αδυναμία να εφαρμοστούν ε, όμορφα ορισμένα πράγματα δημιουργεί πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν κύριε Πελέ τώρα θα σας δώσω δύο λεπτάκια για να μας ε, πείτε τα δικά σας σχόλια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θέλω που δεν είναι λόγο να εξάγω συμπεράσματα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας σήμερα. Ίσα ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας που οργανώνει αυτή την ακρόαση σήμερα. Είδαμε την, την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της δικής σας και ήδη τα αποτελέσματα της δικής μας της έρευνας εν πολύ συνάδουν με τα αποτελέσματα της μελέτης του London Economics. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω με άλλα λόγια κύριε Πρόεδρε. Τώρα, βέβαια εδώ σήμερα άκουσα πολλές και διαφορετικές απόψεις. Η ε, αλήθεια δεν είναι μία. Περιμένουμε όμως εγώ θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να ε, περι, πάρουμε πληροφορίες ε, μέχρι το τέλος του μηνός έχουμε δώσει την προθεσμία αυτή μέχρι το τέλος του μήνα να μας δώσουν πληροφορίες τα κράτη-μέλη για το τι γίνεται στο εσωτερικό τους και μέχρι τον Ιούλιο θα δούμε τι γίνεται και αν άνοιξαν καινούργιοι λογαριασμοί πόσοι λογαριασμοί άνοιξαν μετά την σύσταση Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να αποφασίσουμε ότι δεν λειτουργεί η σύσταση, θα πρέπει να νομοθετήσουμε, να, πρα να πρόκειται για οδηγία κανονισμό. Ε, βέβαια η νομοθεσία ε, έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί κανείς να την επιβάλλει. Ωστόσο το θέμα είναι πώς θα την εφαρμόσει ο καθένας. Αλλά αν νομοθετήσουμε ε, με μια οδηγία, το πούμε, θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να ε, περάσουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία. Θα αργήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε τι, αν τα κράτη-μέλη δηλαδή δεν θέλουν να εφαρμόσουν ορισμένα πράγματα, τα εθνικά τραπεζικά συστήματα, τότε δεν φοβάμαι ότι ούτε και η νομοθεσία θα προχωρήσει γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος, ευχαριστώ που είστε εδώ. Τώρα... να δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές. Εσείς πρώτα από την Οικονομική Επιτροπή. Ναι, νομίζω ότι φάνηκε εδώ από αυτή την ακρόαση ότι είναι υποχρεωτικό να ενεργήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προστατεύσουμε τις πληττόμενες ομάδες. Ε, δεν πρόκειται ε, δεν θέλουμε εδώ τώρα να δούμε μοναχά τι κάνουν Γερμανία ή γιατί λειτουργεί καλύτερα το σύστημα στη Γερμανία. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι βεβαίως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τι θετικές εμπειρίες της Γερμανίας. Αλλά το θέμα δεν είναι να εξάγουμε ή να εφαρμόσουμε ένα εθνικό μοντέλο. Το θέμα είναι να βρούμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο να εφαρμόσουμε. Και για να κλείσω, να αναφερθώ σε μια ηθική πολιτική αρχή, να πω ότι δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε soft law δεδομένων αυτών που προσπαθούμε να προστατεύσουμε αν θέλετε ε, μην ξεχάσουμε να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για φτωχούς ανθρώπους τους οποίους για να προστατεύσουμε πρέπει να έχουμε νομοθεσία που να επιβάλλεται. Η κυρία Γκέιπχαρτ, ε, χαίρομαι που έγινε η ακρόαση αυτή, ε, χαίρομαι που άξιζε που έγινε ακούσαμε διαφορετικές απόψεις είτε εξάγουμε μονοσήματα συμπεράζουμε είτε όχι κύριε Στάιν στην αρχή της παρέμβασής σας είπατε ότι και αυτοί που ασχολούνται με την προστασία του καταναλωτή και αυτοί που ασχολούνται με, την τράπε, με τις τράπεζες συμφώνησαν. Μα συγγνώμη τότε γιατί έγινε στο Κοινοβούλιο αυτή η εντονότατη συζήτηση που έγινε τις τελευταίες μέρες. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι υπάρχει συνένεση εκεί και το ότι η γερμανική κυβέρνηση λέει δεν κάνω τίποτε αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι ξέρει ότι γίνεται γίνονται κάποια πράγματα σε ευρωπαϊκά επίπεδο και δεν θέλει να προτρέξει. Λοιπόν, ή το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα το ότι κάποια πράγματα γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας είναι απαραίτητο να βρεθεί κάποια ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή λύση. Θα ήθελα τώρα όλος ιδιαίτερος να ευχαριστήσω τον κύριο Μιούλερ γιατί ε, είπε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρόκειται μόνο για ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες. Πρόκειται για πάρα πολλές και διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων που έχουν προβλήματα. Δεν είναι μόνο αυτοί που δεν έχουν λεφτά. Δεν είναι μόνο αυτοί που είναι αφαιρέγγοι. Είναι οι φοιτητέ. Οι νέοι αυτοί που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα Εράσμους και πάνε να βιώσουν την Ευρώπη σε άλλη χώρα και ξαφνικά τι βιώνουν, ένα κρύο παγωμένο ντους βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν και αυτές πρόβλημα και μπορεί να χάνουν παραγγελίες επειδή ε, ε, κάποιοι δεν έχουν ε, ε τραπεζικό λογαριασμό. Ευχαριστώ όλους αυτούς που ανέφεραν όλα αυτά τα διαφορετικά παραδείγματα περιέγραψαν όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν ε, θα φτιάξουμε τις εκθέσεις μας, θα τις υποβάλλουμε, θα τις συζητήσουμε και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και στην Επιτροπή ε, Οικονομικών Υποθέσεων θα προχωρήσουμε γρήγορα, ούτω ώστε το αργότερο τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να πάρει μια κάποια απόφαση την οποία να ούτως ώστε η Επιτροπή όταν θα δουλέψει τον Ιούλιο να, έχει, να ξέρει ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για να μπορέσουμε και εμείς λοιπόν να επηρεάσουμε τη δουλειά που θα γίνει στην Κομισιόν. Εμείς ως εκπρόσωποι και άμεσα εκλεγμένοι των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να έχουμε σαφή άποψη την οποία να προωθήσουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και την πολύ καλή ε, ακρόαση. Ευχαριστώ και εγώ λέει ο Πρόεδρος. Uh, we um, Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο εισηγητές και ιδιαίτερα την Evelyn Gebhardt η οποία οργάνωσε την ακρόαση αυτή. Ευχαριστώ όλους αυτούς που έλαβαν μέρος και πριν να κηρύξω τη λήξη της συνεδρίασης να πω ότι Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου θα από τις 3 μέχρι τις 6.30 θα γίνει η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο. Ελπίζω να απίλαυσαν την ακρόαση. Σας ε, τα της ακρόασης θα εμφανιστούν και στην εφημερίδα στο New Sheet της Επιτροπής ε, Εσωτερικής Αγοράς και τέλος ευχαριστώ τους διερμηνείς και εύχομαι σε όλους καλό σας βράδυ.

qua